Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε για σήμερα το πρωί με το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η χρηματοδότηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η συγητής είναι ο κύριος Τόμας Χέντελ και του δίνω ευθύς αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Sehr Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής και Παγκοσμιοποίησης απαιτεί μια προκαταρτική παρατήρηση. Πέρσι ήταν ένα θαυμάσιο μέσο για την αντιμετώπιση της κρίσης για τους εργαζόμενους που έχασαν τις θέσεις τους ε, λόγω της παγκοσμιοποίησης και των επιπτώσεων. Ο στόχος ήταν λοιπόν να ορθολογήσουμε τη λειτουργία αυτού του Ταμείου για να υποστηρίξει αυτούς που έχασαν ή θα χάσουν τις, εργα... τις τους τα επόμενα χρόνια, τον αριθμό των οποίων δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Αλλά οι ανάγκες αυτές διατυπώνονται, προβάλλονται από τους κοινωνικούς εταίρους. Τώρα θέλουμε να ρυθμίσουμε περισσότερο τις λεπτομέρειες, αλλά και να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Η πρώτη παραγράφος αναφέρεται στα μέσα στους πόρους δηλαδή, τους μεμονωμένους, τους οποίους έχουν, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί, στα ποσά τα οποία έχουν διατεθεί για τα εθνικά και τα επιχειρησιακά μέτρα στήριξης. Υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά για τη χρησιμοποίηση αυτών των πόρων σε εθνικό πλαίσιο. Αυτή η έκθεση την οποία θέλουμε να λάβουμε από την Κομισιόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περαιτέρω πορεία του Ταμείου. Δεύτερον, είναι ουσιαστικό να προσπαθήσουμε το Ταμείο αυτό να στοχεύσει ε, πραγματικά στις επιχειρήσεις που χρειάζονται τη στήριξή του. Την προηγούμενη περίοδο επιχειρήσεις ε, εκμεταλλεύτηκαν τους πόρους ε, του ταμείου αυτού χωρίς να έχουν άμεση ανάγκη. Ένα κλασικό παράδειγμα ήταν η κατάσταση του εργοστασίου της μονάδας παραγωγής της Dell στην Ιρλανδία και ζήτησαν 14 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για την κάλυψη, κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων Ε, και είχε δηλώσει η Ντέλ ότι θα κλείσει τη μονάδα αυτή στην Ιρλανδία και θα πάει στην Κίνα. Όμως μερικές εβδομάδες αργότερα η Ντέλ δεν πήγε στην Κίνα, πήγε στην Πολωνία και μετέφερε πολλούς εργαζόμενους από την Ιρλανδία στην Πολωνία. Και τελικά δεν πήρε 14 εκατομμύρια, πήρε 48. Μην ξεχνάμε ότι η Dell δεν είναι ένα φτωχό, μια φτωχή και αδύναμη εταιρεία είναι μια τεράστια πολυεθνική με κεφάλαιο τριών δις. Λοιπόν, πρέπει να φροντίσουμε <clears throat> να μην πηγαίνουν οι πόροι αυτοί σε λάθος χέρια εις βάρος των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Και γι' αυτό η παράγραφος 3 ζητεί ε, την ε, συμμετοχή επιχειρήσεων μόνο σε περίπτωση, σε περίπτωση που ε, προβάλλουν βάσιμα επιχειρήματα για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων αναπλήρωσης. Πρέπει και οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο κοινωνικό κόστος, εάν θέλουν να λάβουν τα ωφέλη του Ταμείου. Τέταρτον, είναι σημαντικό να δοθούν οι πόροι αυτοί για την εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης και ιδιαίτερα σε αδύναμες περιοχές όπου χρειάζεται ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει οι πόροι αυτοί να καλύπτουν ε, περιφέρειες ε, ανάπτυξης, να έχουν στόχους περιφερειακής ανάπτυξης δεδομένου ότι αυτός είναι ο στόχος της ε, χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών μέτρων, των ευρωπαϊκών πόρων. Ε, πέμπτον, το συζητήσαμε και χτες ε, την υποχρεωτική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Είπαμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Η παράγραφος 6 αναφέρεται σε σημεία στα οποία έχουμε ακόμα δυσκολίες, δηλαδή την υλοποίηση σε ένδο, ενδοευρωπαϊκό πλαίσιο όταν επιχειρήσεις μεταφέρονται εντός της ε, επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα θέλουμε να απλοποιηθεί η υποβολή αιτήσεων ε, για την παροχή πόρων ε, όταν πρέπει να γίνουν γρήγορες μετατροπές ε, και χάνονται θέσεις εργασίας αλλά ανοίγουν άλλες ευκαιρίες αλλού. Και έβδομον deutlich Ζητούμε από την Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά το, τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης δεδομένου ότι δεν προβλέπεται άμεση ε, λήξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ε, γι' αυτό λοιπόν ζητούμε την αύξηση του χρηματοδοτικού πλαισίου σημαντικά και να δοθεί έναν, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο αυτό ένας δικός του τίτλος ε, στον προϋπολογισμό. Ένας οικείος τίτλος στον προϋπολογισμό. Αυτά κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάντελ. Η κυρία Χούμπνερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην Ευρώπη μπαίνουμε σε μία περίοδο που η οδηγία για την Βασιλεία θέλει να ενισχυθεί και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα χρήματα ε, που έχουν οι πολίτες μας είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε, σωστά, λέει ο εισηγητή, πρέπει να αισθήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα για την βελτίωση του Ταμείου. Όμως, επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι είναι επίση προφανές ότι αντιμετωπίζουμε διαρθρωτικές τροποποίησεις στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Επιχειρήσεις οι οποίες πήγαιναν καλά πριν από την κρίση, πολύ συχνά σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και είναι λογικό να περιμένουμε ότι νέε θέσει απασχόληση, εφόσον δημιουργηθούν, θα δημιουργηθούν σε νέου τομεί και σε νέε επιχειρήσει. Πρέπει να δούμε τι προσδοκίε των καταναλωτών σε σχέση με νέες αγορές που αναπτύσσονται με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Όλες αυτές είναι αλλαγές που έχουν ξεκινήσει να έχουν ήδη επιπτώσεις στις κοινωνίες μας. Όμως με όλες αυτές τις αλλαγές υπάρχει και μια πρόκληση και μια ευκαιρία μπροστά μας. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα αντιδράσουμε στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες αυτές, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές προκλήσεις των οποίων οι επιπτώσεις δεν θα πρέπει να είναι τέτοιες που να καταστρέψουν τις ευκαιρίες. Είναι σημαντικό λοιπόν σήμερα να εντοπίσουμε και νέες πηγές ανάπτυξης και να επικεντρωθούμε σε αυτές. Περί αυτού θα έπρεπε να πρόκειτο η στρατηγική 2020. Σίγουρα λαμβάνει υπόψη και την βιομηχανική πραγματικότητα της Ευρώπης, δεν είναι μόνο πράσινη. Η στρατηγική αυτή λοιπόν θέλει να συμπεριλάβει και νέα στοιχεία, αλλά και να αλλάξει δια... παλιά μοντέλα και παλιές δομές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα στην απασχόληση που πρέπει να προστατεύσουμε και την απασχόληση που πρέπει να αντικαταστήσουμε με νέα. Και είναι δύσκολο αυτό. Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε πολλή ανάπτυξη και καταλαβαίνουμε ότι μέρος της ανάπτυξης ε, αυτής ε, θα είναι με απόλυτη θέση απασχόλησης αυτών που υπάρχουν σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε πολιτικές και εργαλεία που θα βοηθούσαν την Ευρώπη να μπορέσει να ανταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να έχουμε τις θέσεις απασχόλησης που θέλουμε. Και εδώ έχω αρκετές αμφιβολίες όσον αφορά τα σημεία σας 2, 3 και 6 και ελπίζω να υπάρξει καρποφόρα συζήτηση μεταξύ των εισηγητών, γιατί φοβόμαι ότι με αυτά που λέτε εδώ θα περιορίσουμε τις διευθυντικές αλλαγέ, θα προσφέρουμε μάλλον αρνητικά κίνητρα στι επιχειρήσεις και δεν θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τις δομές αυτές που δεν είναι αρκετά ε, ανταγωνιστικές σήμερα στην Ευρώπη. Εμεί χρειαζόμαστε θέσει απασχόληση που δεν θα χαθούν μεθαύριο όταν θα έχουμε νέε εξελίξει. Η Ευρώπη μπορεί να αναπτυχθεί μόνο όταν έχει ανταγωνιστική βιομηχανία. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας, σαν κύριο θέμα, ότι το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση πρέπει να στηρίζει τις διαφορετικές αλλαγές. Δεν θέλουμε με αυτό να αποφύγουμε διαφορετικές αλλαγές, όχι. Αυτό πρέπει να είναι το κύριο σημείο του θέματος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ποδηματά τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον ε, εισηγητή ε, για το σχέδιο γνωμοδότησης που έχει υποβάλει. Θεωρώ πολύ σωστή την ε, χρονική στιγμή και την πρωτοβουλία για να γίνει μια έκθεση αποτίμησης της χρηματοδότησης και της μέχρι σήμερα λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην ε, παγκοσμιοποίηση με δεδομένο ότι στα δύο χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει από την ε, θέση σε ισχύ του σχετικού ε, κανονισμού έχει καταγραφεί και αυτό επισημαίνεται στο σχέδιο γνωμοδότησης περιορισμένη χρήση αυτού του νέου χρηματοδοτικού μέσου. Η έκθεση της Επιτροπής ως προς την αξιολόγηση της μέχρι σήμερα ανάληψης δράσεων από το Ταμείο νομίζω ότι θα πρέπει και μπορεί να συνοδεύεται από συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία κράτος μέλος ε, με στόχο να αναδειχθούν και να επισημανθούν οι βασικές αιτίες που οδήγησαν στην περιορισμένη χρήση αυτού του σημαντικού χρηματοδοτικού ε, εργαλείου. Ε, ως ο κατεξοχήν λόγος για την περιορισμένη κινητικότητα των πόρων του Ταμείου ε, θεωρείται η ύπαρξη πολύπλοκων διαδικασιών, γεγονός που καθιστά ε, χρονοβόρα και περίπλοκη τη διαδικασία ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην ε, ε, παγκοσμιοποίηση με επιπρόσθετο κόστος για την κρατική μηχανή για το δημόσιο τομέα των κρατικών μελών. Ένα πρώτο βήμα λοιπόν μετά την αξιολόγηση της μέχρι σήμερα λειτουργίας και εφαρμογής του κανονισμού θα ήταν νομίζω η προσπάθεια απλούστευσης ε, των σχετικών διαδικασιών και ταχύτερης ε, διεκπαιρέωσης, ταχύτερης ικανοποίησης των ετοιμάτων ε, ενεργοποίησης. Στο ίδιο πλαίσιο θα μπορούσε να προταθεί και η οριοθέτηση εξ αρχής αρμόδιου εθνικού φορέα σχετικά με την διαχείριση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με τρόπο που να διευκολύνει ε, τόσο την ανάπτυξη τεχνογνωσίας όσο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν ε, στο, ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνδυασμό βεβαίως με τη μεγαλύτερη κινητοποίηση και ενημέρωση ε, των εθνικών αρχών από την πλευρά της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές επιμέρους παρατηρήσεις και επισημάνσεις γύρω από το σχέδιο γνωμοδότησης. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με την πρόταση του εισηγητή στην παράγραφο 2 ε, με την ε, οποία καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση η οποία να προβλέπει τη συμμετοχή επιχειρήσεων κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο οι οποίες καταργούν θέσεις εργασίας και σημείωσαν κέρδη κατά τις προηγούμενες περιόδους ε, εκθέσεων στο συνεπακόλουθο κοινωνικό κόστος της μεταφοράς επιχειρήσεων και άρα κατάργησης θέσεων εργασίας. Νομίζω ότι επί της αρχής ε, είναι μια ε, σωστή πρόταση που θα μπορούσε ασφαλώς να εξειδικευτεί περαιτέρω ε, εστιάζοντας κυρίως στις επιχειρήσεις εκείνες των οποίων η μετεγκατάσταση η αλλαγή έδρας δεν συνδέεται με το ζήτημα της μακροχρόνιας οικονομικής τους βιωσιμότητας αυτό είναι μία επιλογή την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε ή εστιάζοντας σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει κάθε είδους κρατική ή κοινοτική χρηματοδότηση ε, την τελευταία πενταετία πρώτης μετεγκατάστασής τους, ε, για παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ποδηματά. Ο κύριος Χάγκλινγκ παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είχα τη χαρά να εργαστώ πάνω στο θέμα αυτό στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Γενικά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μία διαφορά μεταξύ ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους και τις βοήθειες σε επιχειρήσεις. Πολλές φορές τα δύο αυτά πράγματα μπλέκονται. Ενώ πρέπει να υπάρχει μία διαφοροποίηση. Γενικά η προσέγγιση μας είναι πρώτον να αξιολογήσουμε αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα. Πολύ σωστά και η γνωμοδότηση είναι πολύ σωστή. Τώρα, τα συμπεράσματα που, συνάγει που εξάγει ο εισηγητής είναι ένα διαφορετικό, διαφορετική ιστορία. Αυτό το Ταμείο Αναδιάρθρωσης, το οποίο θα βασίζεται ε, σε μία εισφορά μεταφοράς έδρας, ε, ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, είναι πολλές φορές ε, χρήματα τα οποία έχουν δοθεί από το ταμείο αυτό ε, ε, ενώ δεν έχουμε εξετάσει ακριβώς πού πήγε η επιχείρηση. Λόγω της παγκοσμιοποίησης πρέπει να παρακολουθούμε ακριβώς πού έχει μεταφερθεί η έδρα πριν δίνουμε, δώσουμε πόρους. Αυτό επί του σημείου δύο. Επί του σημείου 3 πρέπει να εξετάσουμε εάν είναι ο ρόλος της Ευρώπης να ε, έχει ένα ταμείο το οποίο υποστηρίζει τις θέσεις αναπλήρωσης. Ε, δεν ξέρω αν αυτό είναι ο ρόλος ακριβώς του ταμείου. Πρέπει να το συζητήσουμε. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων ε, είναι μία δύσκολη υπόθεση και από απόψε τεχνικής υλοποίησης δηλαδή, να συμμετέχουν πάντοτε οι κοινωνικοί εταίροι. Δεν είναι κακή ιδέα, αλλά δύσκολα εφαρμόζεται. Στο σημείο 6, ένα ταμείο το οποίο υποστηρίζει τις ενδοευρωπαϊκές μεταφορές επιχειρήσεων, για μένα αυτό είναι εντελώς αντίθετο με τη βασική ιδέα του ταμείου, με τους βασικούς στόχους δεν μπορώ να υποστηρίξω το σημείο 6 διόλου. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μία εις συζήτηση. Το σημείο 7, όπως είπε και η κυρία Χούμπνερ, η οικονομική πραγματικότητα μάλλον δεν μας επιτρέπει να ε, εμπλουτίσουμε πολύ περισσότερο αυτό το ταμείο. Δεν νομίζω ότι έχουμε περισσότερα χρήματα να ξοδέψουμε για το ταμείο αυτό και να αυξηθούν οι πόροι του. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν πρέπει να κάνουμε μία εις και ενδελεχή συζήτηση με τον εισηγήτη και θα ε, υποβάλω και τροπολογίες τις οποίες θα συζητήσω μαζί του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Χάτον, η κυρία Εστρέτσεκ. Ο κύριος. Ευχαριστώ, καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθώ και εγώ με μεγάλη προσοχή τη συζήτηση και θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω μια διαφορετική προσέγγιση. Ο συνάδελφός μου, κύριος ε, Χαμπλούντ, με κάλυψε σε ορισμένα σημεία, αλλά έχω και εγώ να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Πιστεύω, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής και Παγκοσμιοποίησης ήταν ένα επίμαχο θέμα εξ αρχή. Εν πάση περιπτώσει, δημιουργήθηκε γεννήθηκε και τώρα είναι εν ζωή. Τώρα η πορεία του δείχνει ότι έχουν ληφθεί ορισμένες αποφάσεις για το ταμείο αυτό, το οι οποίες από οικονομικής απόψεως δεν ήταν και πολύ καλές. Ήταν επίμαχες και αντιφατικές. Αυτές οι αποφάσεις δηλαδή που έλαβε το Ταμείο. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι πόροι αυτοί χρηματοδοτούνται από ε, χρήματα φορολογούμενων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όταν μιλάμε για παγκοσμιοποίηση είναι βεβαίως λογικό ορισμένοι να επιβιώσουν και να είναι επιτυχείς, ορισμένες επιχειρήσεις, άλλες να μην, είναι, να μην μπορούν να ανταγωνιστούν και να βουλιάξουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες ε, ζημιώνονται λόγω της παγκοσμιοποίησης. Δεν μπορούμε δηλαδή τεχνικά, να κρατήσουμε εν ζωή επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες. Πρέπει να υποστηρίξουμε επιχειρήσεις που προσφέρουν νέες θέσεις, καινοτομίες, νέα προϊόντα και ούτω καθεξής. Επίσης πρέπει να φροντίσουμε τη σωστή χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Αυτό είναι ε, και δει για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο... Οι, ε, Ευρω... οι Βρετανοί συντηρητικοί θα ζητήσουν μία λεπτομερή αξιολόγηση της έκθεσης αυτής από την Κομισιόν. Ε, θέλουμε η Επιτροπή να μας υποβάλει μία έκθεση λεπτομερή με όλα τα στοιχεία. Τι λεφτά δόθηκαν σε ποιον, για ποιο λόγο, για πόσους εργαζόμενους, τι έγιναν αυτές οι επιχειρήσεις, να έχουμε δηλαδή ε, όλα τα στοιχεία της λειτουργίας και της διάθεσης των πόρων για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την λογική, τη συνετή λειτουργία αυτού του Ταμείου και τη σωστή διάθεση των πόρων. Αυτό το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης υποτίθεται ότι ήταν ένα χρηματοδοτικό κανάλι το οποίο θα λειτουργούσε παράπλευρα με τα ευρωπαϊκά διαστρωτικά ταμεία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω κανάλια, περαιτέρω ο, ο, ο, άλλες, άλλες οδούς ε, χρηματοδότησης. Ε, ε, φτάνουν αυτά τα οποία έχουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Στέσσεκ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Γιόγκερσεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε αυτή, που είναι και η πρώτη ευκαιρία που έχουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, που είναι υπεύθυνε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, να έρθει εδώ και να σας απευθύνει το λόγο. Θέλω λοιπόν να κάνω κάποια σχόλια στις προτάσεις που κάνει ο εισηγητής. Πρώτα απ' όλα θέλουμε επικοδομητική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να είναι έτοιμο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ένα ταμείο το οποίο θέλει να στηρίξει τους ε, ε ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους και όχι για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις. Καμία επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπεριλαμβάνω και την Ιρλανδία. Καμία λοιπόν επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πάρει οικονομική χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία αναφερθήκατε δεν υπήρξε στήριση για τη μετεκατάσταση της επιχείρησης. Ελέξαμε πάρα πολύ καλά κατά πόσο επρόκειτο για μετεκατάσταση θέσεων απασχόλησης. Δεν υπήρχε τέτοια μετεκατάσταση από την Ιρλανδία στην Πολωνία. Τα προϊόντα και η διαδικασία παραγωγής διαφέρουν. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω κύριε Χούμπνερ για αυτό που είπατε για την πρωτοβουλία 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ξεκάθαρα ότι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι ένα από τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε. Αναφέρουμε το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση όσον αφορά τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα γιατί το Ταμείο αυτό πρέπει να στηρίξει αναδυόμενε αγορές η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις και δουλεύουμε σκληρά πάνω σε αυτό για να δούμε πώς μπορούμε να το θέσουμε όντω σε εφαρμογή. Χαίρομαι επίση για τι ιδέε που ακούσαμε όσον αφορά την ανάπτυξη του Ταμείου προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ιδιαίτερα θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τις διαδικασίες που διέπουν την χρήση των κονδυλίων του Ταμείου αυτού. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, βασιζόμαστε στις 22 περιπτώσεις όπου εδώ έχουμε ένα πλήρη κύκλο χρηματοδότησης. Ο μέσος ε, όρος χρόνου από τη στιγμή όπου η Επιτροπή έχει την πλήρη ενημέρωση από τα κράτη-μέλη μέχρι τη στιγμή της πληρωμής από την Επιτροπή στο λογαριασμό του θησαυροφυλακίου του, κρατού, του κράτους μέλους έχουμε 225 μέρες κατά μέσο όρο. Εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε μειώσει τις δικές μας διαδικασίες. Έχουμε συγχωνεύσει δύο διαδικασίες σε μία και έτσι έχουμε κερδίσει 22 μέρες από τις 225. Αυτή την εποχή προσπαθούμε να δούμε μήπως μπορούμε να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο κατά 40-45 μέρες από τη διαδικασία σε σχέση με την πληρωμή των πιστώσεων αλλά αυτό απαιτεί αναθεώρηση των δημοσιονομικών διαδικασιών που εφαρμόζει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι θα πρέπει όμως να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό και σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο ε, έχει τα κονδυλιά του το ταμείο αυτό πρέπει να υπάρξει επίσημη ε, έγκριση από τη Δημοσιονομική Αρχή, που σημαίνει και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα πρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε οι διαδικασίες να λάβουν χώρα σωστά από τις δύο αρχές που είναι υπεύθυνε για τον προπολογισμό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη διαδικασία εκτός αν αλλάξουμε και τον κανονισμό και τις δημοσιονομικές προοπτικές και την διοργανική συμφωνία. Νομίζω ότι δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν έρχομαι τώρα στο δεύτερο σημείο μου, που είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος πότε μπορεί να γίνει πρόταση για θεωρημένο κανονισμό. Φυσικά υπάρχει ένα ραντεβού για του χρόνου, γιατί του χρόνου είναι και η τελική χρονιά όσον αφορά τις παρεκκλήσεις εξαιτία τη κρίση και πρέπει να ληφθεί απόφαση για το κατά πόσο θα συνεχιστεί η παρέκκληση ή θα προτείνουμε κάτι διαφορετικό. Όμω υπάρχει και σύνδεση με τη συζήτηση που γίνεται για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και για την ε, δομή του επόμενου προπολογισμού. Ο Αρμόδιος Επίτροπος στην Σουηδία είπε την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς αυτό που έχετε και εσείς στο σημείο 7 στις προτάσεις σας. Ότι δηλαδή πρέπει να δημιουργηθεί μια γραμμή στον προπολογισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στις δημοσιονομικές προοπτικές, ώστε να βρεθεί το Ταμείο αυτό επί ίσης ώρες με άλλα ε, δημοσιονομικά μέσα. Η απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα πάντως. Ε, θα το δούμε αργότερα. Και ένα τελευταίο σημείο που έχει να κάνει με το δικό σας σημείο 1, όπου χαιρόμαστε πολύ που κάνετε έκκληση για περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη διαφάνεια και καλύτερα στατιστικά δεδομένα για το Ταμείο. Ετοιμάζουμε τώρα την ετήσια έκθεση για το 2010 που θα είναι έτοιμη σε ένα μήνα περίπου. Και για πρώτη φορά προτείνουμε με έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγκεντρώνουμε όλα τα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε σε μία βάση, οπότε θα υπάρχει ένα παράτημα στατιστικό που θα δείχνει με περισσότερες λεπτομέρειες την φύση των αιτήσεων, ε, αναφύλλο, αναηλικία, ανακλάδο που στηρίζουμε, τον αριθμό των ανθρώπων που στηρίζουμε με τα διάφορα μέτρα κλπ. Αυτή είναι μόνο η αρχή μιας προσπάθειας που γίνεται να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Συμβούλιο και στους ενδιαφερόμενους από το κοινό. Στηρίζουμε την ιδέα ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οργανώσει συναντήσεις με εκπροσώπους από όλες τις χώρες μέλη σε τακτική βάση, δύο φορές το χρόνο δηλαδή. Έχουμε οργανώσει και σεμινάρια για να εξηγήσουμε πώς ε, δουλεύει και πώς ερμηνεύεται ο κανονισμός. Στις συναντήσεις αυτές και στις επαφές αυτές έχουμε ανταλλαγή απόψεων και μεταξύ των χρηστών του Ταμείου, έτσι ώστε να μπορεί ο ένας να εμπνευστεί από τις ιδέες ε, κάποιου άλλου. Προσδοκώ ε, συνέχιση των επαφών μεταξύ μας και έχω σημειώσει ό,τι προτάσεις κάνατε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιόγκερσεν. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Χάντελ, για να κλείσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τις παρατηρήσεις σας. Θα διαμορφώσουμε λοιπόν ένα σχήμα συνεργασίας για να οριστικοποιήσουμε τη γνωμοδότηση και θα μιλήσω και με την Επιτροπή βεβαίω με την Κομισιόν. Είχαμε ήδη χτες την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων. Πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να συζητήσουμε ε, την περίπτωση μιας επιχείρησης που λόγω αναδιάρθρωσης δεν είναι πια ανταγωνιστικό. Πρέπει λοιπόν το Ταμείο να βοηθήσει τους εργαζόμενους που θα χάσουν ή έχασαν τις θέσεις εργασίας, όχι την επιχείρηση. Τώρα, εάν η επιχείρηση αυτή επεκτείνεται και μεταφέρει τις δραστηριότητες της και ανοίγει μια καινούρια μονάδα παραγωγής σε μια άλλη ε, έδρα. Μεταφέρει δηλαδή την έδρα της ή ανοίγει μια καινούρια μονάδα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εάν σε αυτή την περίπτωση όπου η επιχείρηση δεν κλείνει δεν χρεοκοπεί αλλά μεταφέρει την έδρα της αλλού αν έχει το δικαίωμα το Ταμείο να υποστηρίξει τους εργαζόμενους, δεδομένου ότι πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου τα χρήματα των φορολογούμενων. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι λογικό μια επιχείρηση η οποία είναι κερδοφόρα, παρόλο που έχει μεταφέρει την έδρα της και κερδίζει απλώς αλλού, σε άλλη επικράτεια. Δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να υποστηρίξουμε μια την επιχείρηση αυτή με πόρους του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Αυτό δεν είναι παράλογο. Αλλά εάν μια επιχείρηση η οποία κλείνει διότι δεν είναι ανταγωνιστική, διότι δεν μπορεί να σταθεί στο παγκόσμιο περιβάλλον και χάνουν τις θέσεις εργασίας τους άνθρωποι, τότε πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Το ανθρώπινο δυναμικό αυτή τη διαφορά πρέπει να την τονίσουμε. Σύμφωνο και είμαι ανοιχτός, μπορείτε να, να συζητήσετε μαζί μου για οποιοδήποτε άλλο θέμα και περιμένω τα, τα σχόλιά σας για να τα εντάξω. Ευχαριστούμε πολύ. Η ημερομηνία προθεσμία πιο σωστά για την κατάσταση τροπολογιών είναι 8 Ιουνίου. 28 Ιουνίου θα συζητήσουμε. Θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας στις 28 Ιουνίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών θα λάβει χώρα στις 14 Ιουλίου 2010. Κλείνει λοιπόν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και περνάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Το λόγο έχει η εισηγήτρια η κυρία Πιετικάινεν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η προστασία του καταναλωτή καλύπτεται από τέσσερις οδηγίες αυτή τη στιγμή που είναι όλες οδηγίες τύπου ελάχιστης εναρμόνισης. Και αυτό σημαίνει ότι όταν υπάρχουν προβλήματα με την εθνική νομοθεσία είτε πρόκειται για συμβατικό δίκαιο είτε για υψηλότερα επίπεδα αυτά καλύπτονται από την εθνική νομοθεσία που διαφέρει από μέρος σε μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, απόπειρα της Επιτροπής αυτή τη φορά και από τα κράτη ήταν ε, διαφορετική, διότι ε, λάμβανε υπόψη την, ε, ότι η ανάγκη για υψηλότερη προστασία μπορεί να καλυφθεί σε εθνικό επίπεδο. Τώρα η Κομισιόν προτείνει να συνδυαστούν αυτές οι τέσσερις οδηγίες και να υπάρξει εναρμόνιση. Τι συμβαίνει τώρα. Προσπαθεί να μετατρέψει τη με εναρμόνιση σε πλήρη εναρμόνιση και αυτό προκαλεί πολύ σοβαρά προβλήματα σε τεχνικό επίπεδο αλλά και επί της ουσίας. Καταρχήν, να σας μιλήσω για το νέο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που ισχύει μετά από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Διασφαλίζει ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και θα πρέπει τουλάχιστον να τεθεί αυτό το ερώτημα, κατά πόσο δηλαδή η πλήρης εναρμόνιση αυτών των αρχών είναι κατά του χάρτη των θεμελιδών δικαιωμάτων και του στόχου ενός υψηλότερου επίπεδου προστασίας του καταναλωτή. Κατά δεύτερο λόγο, η στρατηγική ΕΕ για το 2020 περιλαμβάνει το στόχο της υψηλής ποιότητας των προϊόντων καθώς και περιβαλλοντικούς στόχους όσον αφορά τα, βιώσιμα σχήματα παραγωγής. Ε, ε, μέσω αυτής εδώ της ε, πρότασης, αντί να αυξάνεται η προστασία του καταναλωτή, μειώνεται. Με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη ποιότητα των προϊόντων, αλλά και τη χαμηλότερη προστασία του περιβάλλοντος. Είναι προβληματικό λοιπόν αυτό το θέμα. Τέταρτο προβληματικό θέμα είναι το εθνικό συμβατικό δίκαιο. Γιατί ξέρετε ότι οποιοδήποτε μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο ή ένα απλό μπουκάλι νερό είναι πολύ διαφορετική υπόθεση. Και το εθνικό συμβατικό δίκαιο είναι περίπλοκο και υπήρξε μια πολύ περίπλοκη συζήτηση για να δούμε πώς θα ενταχθούν οι εθνικές νομοθεσίες σε αυτή την πλήρη εναρμόνιση. Κάτι πολύ θετικό το οποίο υποστηρίζω στην πρόταση της Επιτροπής είναι ότι θα πρέπει να αυξηθούν η διασυνοριακή αγορά προϊόντων αλλά και το οι ηλεκτρονικές αγορές. Τώρα, αυτό που είναι αμφισβητήσιμο είναι κατά πόσο η εναρμόνιση των, των δικαιωμάτων των καταναλωτών θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Αν συγκρίνουμε το σύστημα με αυτό τον ΕΠΑ, υπάρχουν διαφορές πολύ σημαντικές όσον αφορά τα επίπεδα προστασίας του καταναλωτή στις διάφορες πολιτείες. Και παρόλα αυτά η εσωτερική τους αγορά λειτουργεί πολύ καλύτερα. Επιπλέον, ορισμένοι πολιτές στο e-commerce, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, λένε ότι προσπαθούν να λύσουν αυτές τις διαφορές ε, ακολουθώντας τη μέθοδο του καλύτερου επίπεδου, δηλαδή προσφέρουν στον καταναλωτή την καλύτερη πρακτική κάθε φορά, το καλύτερο μοντέλο. Δεν το θεώρησαν πρόβλημα. Όμως δεν έχουν δει και αντίστοιχη αύξηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τώρα, Όσον αφορά το θέμα της γλώσσας, της εμπιστοσύνης, αλλά και της εμπιστοσύνης στο σύστημα πληρωμών έχουμε πρόβλημα και πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να δουλέψουμε για την αρμόνιση του συστήματος πληρωμών, που πράγμα που εκκρεμεί και μάλιστα φαντάζομαι ότι το ψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή θα μπορούσε να αυξήσει την ε, εμπιστοσύνη του καταναλωτή και αντί να έχουμε αυτή τη συμβαστική προσέγγιση εδώ. Αυτή η ε, πρόταση λοιπόν, ε, μάλλον όλοι αυτοί οι λόγοι με οδηγούν στο να πω ότι δεν πρέπει να εναρμονίσουμε τους κανόνες προστασίας του καταναλωτή. Όμως, ο ίδιος ο στόχος είναι καλός και αποτελεσματικός με την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει προς το ψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Δεν είμαι λοιπόν κατά της πλήρους εναρμόνισης, αλλά είμαι κατά της μεθόδου και του επίπεδου στο οποίο φτάνει αυτή η πρόταση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να εναρμονίσουμε μόνο το πρώτο κεφάλαιο. Ορολογία δηλαδή, πώς ορίζουμε τα διάφορα στοιχεία. Επιστροφή των αγαθών και ένα σωρό ίσονο σημασία θέματα, αλλά όχι όλα αυτά τα δύσκολα σημεία. Και ακόμα δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Καταρχήν για τις περαιτέρω εξελίξεις είναι λυπηρό που η Κομισιόν δεν μπόρεσε σε αυτή τη φάση να προβλέψει την ανάπτυξη των αγαθών καλύτερα. Δηλαδή έχουμε όλο ένα και περισσότερο τέτοια αγαθά όπου συνδυάζουμε ένα αγαθό και μια υπηρεσία, δηλαδή υλικό και άϊλο προϊόν. Έχουμε ας πούμε ένα λογισμικό, ένα τηλέφωνο και έχουμε και τη μουσική που έρχεται με το τηλέφωνο. Μπορεί ο καταναλωτής ας πούμε να είναι, να είναι ευχαριστημένος με το λογισμικό αλλά να μην είναι ικανοποιημένος με τη μουσική γιατί δεν έχεις ας νέα μουσική για ένα χρόνο. Αυτό είναι λάτωμα του προϊόντος ή όχι. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αλλάξουμε τον όρο εκεί και να μιλάμε όχι μόνο για υλικά αλλά και για άλλα αγαθά. Κάτι ακόμα που θέλουμε να λάβει υπόψη η Επιτροπή είναι ότι χρειαζόμαστε εναλλακτικέ επίλυσης διαφορών σε εθνικό επίπεδο και σε ε, ε διεθνές επίπεδο. Τώρα το πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει αυτό μπορεί να είναι δύο χρόνια ή δέκα χρόνια γιατί δεν είναι λογικό για τον παραγωγό να περιμένει ότι αυτό το στυλό θα διαρκέσει περισσότερο από δύο χρόνια ας πούμε αλλά για άλλο είδους προϊόντα μπορεί να περιμένουμε μεγαλύτερη διάρκεια αν είναι καλοφτιαγμένα και να υπάρξει αυτή η προσαρμογή και να είναι δίκαιη για τον πολιτή και για τον καταναλωτή χρειάζεται αυτού του είδους η μέθοδος επίλυσης διαφορών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι λογικό να αναμένει κανείς. Και έρχομαι έτσι στο θέμα που ορίζεται πολύ διαφορετικά από τα διάφορα κράτη σε σχέση με το πιο τι είναι ελάττωμα και ποιος είναι υπεύθυνο για τα ελαττώματα ενός προϊόντος. Επίσης, το θέμα της ρύθμισης των προϊόντων ε, που ορίζονται στις διάφορες οδηγίες είναι πάρα πολύ θετικό. Το μόνο πρόβλημα είναι όταν έχουμε μικρά μικροπροϊόντα τα οποία δεν εμπίπτουν στο φάσμα των άλλων οδηγιών ή ας πούμε πιστώσεις που μπορεί να πάρει κανείς για ένα κινητό τηλέφωνο οι ασφαλίσεις που συνοδεύουν την πώληση του προϊόντος ή άλλα ζητήματα. Όλα αυτά μπορεί να χρειαστεί να ρυθμιστούν στο μέλλον μέσω της οδηγίας που αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή και της οδηγίας του κανονισμού που αφορά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τέσσερις έχουν ζητήσει το λόγο. Και έχουμε και την Επιτροπή και μετά πρέπει στις 10 ε, να ψηφίσουμε, έτσι. Πέντε έχω ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ να είσαστε σύντομοι. σας Πρεσέδο πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Η εκθεσή της είναι καλή, πιστεύω, συμφωνώ και βασίστε στις συζητήσεις που είχαμε νωρίτερα. Θέλει να συμπληρώσει τις ε, διάφορες πτυχές που υπάρχουν. Και εγώ τρία πράγματα έχω να πω εδώ. Πρώτον, για την ίδια τη φύση της οδηγίας όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεύτερον, όσον αφορά τις επιπτώσεις στη... στο δημοσιονομικό τομέα. Και τρίτον, την μεταχείριση που έχουν οι καταναλωτέ οι καταναλωτές όσον αφορά τα δημοσιονομικά προϊόντα. Λοιπόν, δικαιώματα των καταναλωτών είναι ο τίτλος. Η οδηγία όμως συνδυάζει τέσσερις οδηγίες χωρίς όμως να προσφέρει ένα οριζόντιο μέσο για την προστασία των καταναλωτών. Και γιατί, γιατί θέλει να προωθήσει την εσωτερική αγορά. Αν θέλουμε λοιπόν οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, τότε τα δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να είναι και ο κατά προτεραιότητα στόχος μας και βέβαια προστατεύοντα τα δικαιώματα των καταναλωτών, προωθούμε και την εσωτερική αγορά. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι όταν μιλάμε για την αναρμόνιση. Η αναρμόνιση είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο. Δεν είναι πανάκια για τα διάφορα επίπεδα. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν μία απλή αναρμόνιση μπορεί να περιορίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών και στον τομέα της εσωτερικής αγοράς που υπάρχουν διάφορες νομοθεσίες, ο περιορισμός των δικαιωμάτων ε, των καταναλωτών περιορίζει και την εσωτερική αγορά. Άρα λοιπόν όταν αποδυναμώνονται τα δικαιώματα των καταναλωτών, αυτό που κάνουμε είναι ο κολεύουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πάντως η πρόταση Μόντι είναι ξεκάθαρη από αυτού. Όταν λοιπόν μιλάμε για πλήρη αναρμόνιση, πρέπει να ελέγξουμε τα πράγματα. Μόνο όταν είναι αναγκαίο αυτό για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Μόνο τότε να γίνεται. Και πρέπει επίσης να επιμείνουμε τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πιο ευνοϊκούς όρους προστασίας των καταναλωτών. Δεύτερο τώρα, δημοσιονομικές αγορές. Αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ είναι μια οριζόντια οδηγία ή όχι. Αν ήταν οριζόντια έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και τις δημοσιονομικέ αγορές. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κάτι οριζόντιο, αλλά από την άλλη μεριά συμφωνώ για το ότι οι δημοσιονομικές υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερη φύση και ότι οι υπηρεσίες αυτές και τα προϊόντα αυτά είναι διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Οπότε, να μιλάμε για μερική παρέκκληση δεν μου φαίνεται σωστό. Το καλύτερο θα ήταν να βάλουμε δύο ρήτρε. Μία ειδική ρήτρα πρώτον που να λέει ότι οποιαδήποτε διάταξη όταν πρόκειται για ειδικέ περιπτώσεις στις δημοσιονομικές υπηρεσίες έχει διαφορετική μεταχείριση. Και δεύτερον, μια άλλη ρήτρα η οποία να είναι να μιλάει για τις πιο ευνοϊκές διατάξεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί αλλιώς πλήττονται τα δικαιώματα των καταναλωτών και άρα και η ίδια η λειτουργία Τη εσωτερική αγοράς. Υπάρχουν τώρα και κάποιε πτυχές οι οποίες αναφέρονται, ειδικέ πτυχές της οδηγία. Όπως η απαγόρευση των πωλήσεων όταν δεν έχουν ζητηθεί αυτές. Πώς η απαγόρευση αυτή επηρεάζει περιπτώσεις όπως είναι τα συνταξιδοτικά συστήματα όπου επιχειρηματίε προτείνουν υπαλλήλου άρρητα και πώς γίνεται η ανανέωση των συμβάσεων ε, ασφάλισης που πάλι γίνονται άρρητα. Τέλος, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προχωρήσουμε και να έχουμε μία χάρτα των ε, δικαιωμάτων των καταναλωτών, γιατί έτσι θα απλοποιούσαμε τα πράγματα και θα προθούσαμε καλύτερη ενημέρωση για τον καταναλωτή. Θα αποφεύγαμε επίσης ανεύθυνη δανειοδότηση και θα συμπεριλαμβάναμε και τις βέλτιστες πρακτικές των ε, κρατών μελών. Θα διευκολύναμε επίσης τις διάφορες συμβάσει, τα δημοσιονομικά μήτρωα και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και ετησίω μία έκθεση για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι όλα αυτά πράγματα τα οποία έχουν μείνει σε κρεμότητα αλλά μόνο τότε θα μπορούσαν πραγματικά να μιλάμε για μια οδηγία που προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σμιτ τώρα παρακαλώ σύντομο όμω, γιατί στι 10 θέλω να ψηφίσουμε. you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν κατάλαβα την τελευταία φάση που, ε, φράση που είπατε. Φαντάζομαι πω είπατε ότι πρέπει να είμαστε σύντομοι. Ωραία, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, την εισηγήτρια για καλή συνεργασία, αλλά πιστεύω πω είναι κρίμα που φαίνεται να έχουμε εγκαταλείψει την ιδέα της πλήρους εναρμόνισης. Φιλόδοξία με αυτήν την αναθεώρηση θα έπρεπε να είναι να επιτύχουμε έναν υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεγάλο επίτευγμα αν το μόνο που θα κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μία και μόνη οδηγία από τις τέσσερις που ίσχυαν μέχρι στιγμής και νομίζω ότι στόχος θα πρέπει να είναι τελικά η πλήρης εναρμόνιση. Σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Σάντσες Πρεζέντο για μια οριζόντια προσέγγιση, αλλά και σκεφτόμενοι σε σχέση με τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πιστεύω πως είναι πολύ σωστό το ότι φύγεται αυτό το θέμα η οδηγία που αφορά τις ε, πιστώσεις για τους καταναλωτές υποκλεί δάνεια για λιγότερο από 200 ευρώ. Θα πρέπει να το καταστήσουμε σαφές ότι τα δάνεια για λιγότερα από 200 ευρώ θα πρέπει να καλυφθούν από τούτη την οδηγία. Το πρόβλημα όμως που δημιουργείται με αυτά τα δάνεια μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων ε, είναι μεγάλο γιατί μπορεί να φτάσουν και στο 1000% επιτόκιο και μπορεί να είναι πολύ προβληματικά. Συνήθως ε, πρόκειται για πολύ νέους οι οποίοι παγιδεύονται μέσα σε τοκογλυφικές καταστάσεις με, με ε, πολύ ψηλά επιτόκια και χρειάζεται τελικά να πληρώσουν ε, αντί για 200-400 ευρώ. Είναι πολύ δραματική κατάσταση. Να θίξω λοιπόν και ένα πολύ επίμαχο θέμα. Θα πρέπει να δούμε μια αναφορά σε μια συλλογική διόρθωση, διότι αποκατάσταση γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ ε, θετικό για καταναλωτές που αγοράζουν ε, στο εξωτερικό γιατί κάτι τέτοιο θα αύξανε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα διευκόλυνε τη δυνατότητά τους να κάνουν ε, να, να, να κάνουν σοβαρές αγορές αλλά και μικρά ποσά. Εγώ πιστεύω λοιπόν πω όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο, φάσμα, στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, ιδιαίτερα εφόσον υπάρχει αύξηση αυτών των αγαθών και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών. Και επίση συμφωνώ για τη δήλωση που αφορά εθνικές, το εθνικό συμβατικό δίκαιο. Σας ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Ο Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Οι πράσινοι συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της εισηγήτριας. Να προσθέσω ότι συμφωνούμε και με τα όσα είπε ο Λεσμίτ για την συλλογική προσφυγή και πρέπει αυτό να μπει εδώ αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχουν παρά μόνο δύο τροπολογίες. Υπάρχει μια ολόκληρη αιτιολογική, ε, αιτιολογία μάλλον που θα δικαιολογούσε πολύ περισσότερες ε, τροπολογίες και ήθελα να θέσω την ερώτηση στην ε, εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριο Φόξ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα μου υποστηρίζει την μείωση του φόρτου προς τις εταιρείες που θέλουν να λειτουργούν διασυνοριακά και να αυξήσει την προστασία του καταναλωτή. Ε, συμφωνούμε με την ανησυχία της Πιέτη Κάναν ότι η πλήρης εναρμόνιση των δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της προστασίας του καταναλωτή. Π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να... να να επιστρέψουν ε, και να απορρίψουν τα προϊόντα και ίσως αυτό θα έπρεπε να διευρυνθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και η εγγύηση που δίνουν συνήθως για δύο χρόνια δεν είναι επαρκής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι έξι χρόνια η εγγύηση ε, και δεν θέλουμε αυτό να περιοριστεί. Δηλαδή δεν συμμεριζόμαστε την άποψη για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αλλά επειδή είναι ειδικέ υπηρεσίες πιστεύουμε πως θα πρέπει να μείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Φόξ. Η κυρία Στήλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή ως μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Θα το συζητήσουμε πολύ σύντομα ή το απόγευμα ή αύριο το πρωί. Όσον αφορά τώρα την ε, εναρμόνιση, το θέμα είναι να μην μειώσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, τουλάχιστον τα, ε, τους ψηφοφόρους τους οποίους αντιπροσωπεύω εγώ στη Σκωτία, τους καταναλωτές, σε αυτούς μειώνονται τα δικαιώματα. Υπάρχουν όμως ε, διαφορές ως μεταξύ Σκωτίας και Αγγλίας και μεταξύ άλλων κρατών μελών. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω την εισηγήτρια μήπως πρέπει για την οδηγία δικαιωμάτων των καταναλωτών να επιστρέψουμε πίσω και να ξανασχεδιάσουμε την οδηγία αυτή από το μηδέν. Ευχαριστούμε. η κυρία Πιτικάνα να κλείσει τη συζήτηση πάρα πολύ σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω, θα λάβω υπόψη μου όλα τα σχόλια. Δεν υπάρχουν άλλες τροπολογίες. Γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε με την εναρμόνιση και ότι θα αναλάβω τη συλλογική διόρθωση στην έκθεσή μου εάν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Οπότε, ή θα προχωρήσουμε με την ορολογία της εναρμόνισης ή θα επιστρέψουμε πίσω στο σχεδιαστήριο Να μην προχωρήσουμε όμως με, ένα δούριο ύπο και δημιουργήσουμε προβλήματα και στις δύο πλευρές, εταιρείες και καταναλωτές. Ευχαριστούμε πολύ. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 8 Ιουνίου. Στις 28 ε, θα το συζητήσουμε, στις 13 θα ψηφίσουμε στις 27 στην εσωτερική αγορά και στην Ολομέλεια στην πρώτη σύνοδο του Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί. Αυτά. Για να ξέρετε, εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση και περνάμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ για την πειθαρχία που επιδείξατε. Right, uh, hello everybody. Can... Λοιπόν, θα ψηφίσουμε τώρα. Να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να έχετε τις κάρτες σας. Ελπίζω να έχετε όλες σας τις κάρτες sure της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Is that the right way for that? Was that...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 Uh, λοιπόν, μπορούμε παρακαλώ να κάνουμε μια δοκιμή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με τις κάρτες σας. Να κάνουμε μια δοκιμή παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε κάτι, ό,τι θέλετε. Θέλουμε να δούμε πόσοι ψηφίζουν. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ, μία δοκιμαστική ψηφοφορία. Ωραία, ωραία. Right, δεν έχουμε λοιπόν παραπάνω κάρτες από ό,τι πρέπει, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην κανονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε καταρχάς το σχέδιο γνωμοδότησης του Βέρνερ Λάγκεν για, την αγορέ για τις αγορές παραγόγων. Λοιπόν, συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Παρά, ε, τροπολογία 84 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι παράγραφος 1α υπέρ παρακαλώ του πρώτου τμήματος 84 κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα είναι το υπόλοιπο του κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά πιστεύω ότι καλύπτεται σε άλλο σημείο. Ωραία. Προχωρούμε στο 84. Τροπολογία 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. καταπίπτουν 86-87 συμβιβαστική 10 σε δύο τμήματα κύριε Κάμπεν ναι, έχουμε μια προφορική τροπολογία να υποβάλουμε για το δεύτερο τμήμα της ψηφοφορίας για την συμβιβαστική 10. Θέλουμε να αφαιρεθεί η λέξη «κύριος» και αν η λέξη «κύριος» αφαιρεθεί θα μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε το δεύτερο κομμάτι της ε, τροπολογίας, γιατί γνωρίζουμε ότι το θέμα της ρευστότητας είναι ένα από τα πιο σημαντικά, μια από τις προκλήσεις, άρα νομίζω πως είναι αρκετά ευρύς ο συμβιβασμός. Αντίθετα, το να πούμε πως είναι εκεί το κύριο θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη, ε, θα ήταν κάπως προβληματικό. Αν όλοι συμφωνούν, μπορούμε, να αυτή η λέξη, να συμφωνήσουμε. Ο κύριος Λάγκεν. Συγγνώμη. Αν συμφωνεί η, ε, η κυρία Μπόλτσα που υπέβαλε την τροπολογία, τότε συμφωνεί και ο, και εισηγητής να, δια, διαλυθεί, ε, ε, συγγνώμη, να διαγραφεί η λέξη principal. Ναι. Συμφωνώ διότι επειδή δεν είναι όλοι δεν, η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ε, η αγγλική για όλους. Είμαι υπέρ της διαγραφής της λέξης principal στο δεύτερο τμήμα. Ε, οπωσδήποτε τα δικά σας αγγλικά είναι καλύτερα από τα δικά μου γαλλικά. Οπότε λοιπόν διαγράφεται η λέξη. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της συμβαστικής 10 υπέρ. Κατά, αποχές. Δεκτό το δεύτερο με τη διαγραφή του principal υπέρ κατά άποχες δεκτό ε, χωρίς τη λέξη principal ε, τροπολογία 100 100 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 102 υπέρ κατά άποχες Νομίζω ότι πέρασε, ότι έγινε δεκτή. Θα παρακαλώ να ελέγξουμε την 102. Ψηφίσατε. Ε, έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 103 απεσύρθη 104 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι ε, απερίφθη να ελέγξουμε παρακαλώ παρακαλώ ψηφίστε 104 ψηφίσατε όλοι Έληξε η ψηφοφορία. Απερίφθη. Οπότε, επανερχόμαστε στο αρχικό κείμενο ψηφίζουμε υπέρ του αρχικού κειμένου κατά αποχές δεκτό. 105 υπέρ ε, κατά αποχές και πάλι δεν είμαι σίγουρη. 105 παρακαλώ να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. 105. Ψηφίσατε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες Δεκτή. 106. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή πηγαίνουμε στην 116 υπέρ κατά αποχές δεκτή 117 υπέρ κατά αποχές δεκτή 118 υπέρ κατά Αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη. Παρακαλώ να ελέγξουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία 118. Ψηφίσατε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο παραγράφου 5. Υπέρ κατά δεκτό. 119 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 120 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 121 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σίγουρο. Παρακαλώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά 121. 121. Ψηφίσατε όλοι. Του. Α. Απερίφθη η 121. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω Έγινε δεκτή. Συμβιβαστική 12. Ένα, είναι ένα τμήμα. Ωραία. Είναι ενιαία η συμβιβαστική 12. Δεν χωρίζεται. Λιπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 190 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται η συμβιβαστική 13 υπέρ κατά δεκτή 138 υπέρ κατά αποχές δεκτή 139 ε, έχει αποσυρθεί 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πηγαίνουμε στην 150 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 152 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 15 που έχει μια προσθήκη υπέρ κατά αποχές δεκτή 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε διότι περιλαμβάνεται στη συμβαστική 9 Α, εμφανίζεται δύο φορές στον κατάλογο, αλλά ο εισηγητής την μετακίνησε στη συμβαστική 9. Ωραία. 166 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 167 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 168 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 169 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 172 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική 16, C16, σε δύο τμήματα. Νομίζω. Το πρώτο τμήμα του, της συμβαστικής 16, υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα. Έχουμε δύο εναλλακτικέ λύσεις. Έχουμε μια προφορική τροπολογία από τους σοσιαλδημοκράτες να αντικατασταθεί το τέλος της δεύτερης πρότασης με μια διαφορετική διατύπωση. Αυτό που θα κάνω είναι καταρχάς να ψηφίσουμε το πρωτότυπο δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ του αρχικού δεύτερου τμήματος, υπέρ κατά αποχές, δεκτό. Τώρα Αρχικά το τρίτο τμήμα ήταν προσθήκη. Ας ψηφίσουμε το, το, το τρίτο τμήμα ως προσθήκη Υπέρ, κατά, αποχές. Δεκτό. Ως προσθήκη λοιπόν και όχι ως κείμενο αντικατάστασης. Οπότε στην Ολομέλεια θα τα τακτοποιήσουμε τα τμήματα. 181 ε, υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. 182 υπέρ κατά αποχές δεκτή 183 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβιβαστική C17α υπέρ κατά αποχές δεκτή Προχωράμε στο C18 στο κάτω μέρος της σελίδας υπέρ κατά αποχές δεκτή και στην 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 208 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτό 209 υπέρ κατά αποχές δεκτή 210 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές δεκτή δεν, δεν βρίσκω πουθενά γιατί να καταπίπτει του 2.11 δεν έχω κανένα σημείωμα που να λέει ότι ε, διαδικαστικό. Στο δικό μου κατάλογο λέει ότι καταπίπτει εάν η συμβιβαστική 19 περάσει. Δεδομένου ότι η συμβαστική 18 καλύπτει το 210 με το 214. Οπότε όλη η ιδέα του συμβιβασμού ήταν το CDS ε, trading. Και οι τέσσερις αυτές αναφέρονται στο CDS. Ο εισηγητής κατά τη δική μου αντίληψη δεν καλύπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Αναφέρεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η πρόεδρος. Εντάξει, θα ψηφιστεί ως προσθήκη. Εφόσον δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια. Θα το ξεκαθαρίσουμε στην Ολομέλεια. Μόλις ψηφίσαμε την 211 και έγινε δεκτή. προχωρούμε στη 212. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 213 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 214 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 215 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 216 υπέρ, κατά, άποχες, Παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία 216. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 217. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική C19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δε... Α, συγγνώμη. Ε, στην επόμενη σελίδα... 200... Ε, Επιτροπή Ανάπτυξης ΔΕΒΕ 6 υπέρ, κατά Κα, κανένας δεν ψηφίζει για να δούμε είναι η παράγραφος 6 της ΔΕΒΕ Ε, παρέμβαση του εισηγητή χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Δεν ακούμε. Η πρόεδρος, ο, εισηγη, ο εισηγητής πιστεύει ότι ε, αυτή η παράγραφος καλύφθηκε ε, από τη συμβιβαστική και απερίφθη. Ίσως να ψηφίσουμε, να την καταψηφίσουμε. Λοιπόν, παράγραφος 6. Πρόεδρος, διαδικαστικό, διαδικαστικό. Λέει στις σημειώσεις μου ότι το 231 μέχρι 237 και η ΔΕΒΕ 236 καλύπτονται από τη συμβιβαστική και δεν πρέπει να ψηφιστούν. Ναι, λέει η πρόεδρος, εντάξει. Έγινε μια αλλαγή την τελευταία στιγμή που δεν υπάρχει στον κατάλογό μου. Και ο εισηγητής πιστεύει ότι έχει καλυφθεί αυτή η τροπολογία, οπότε έληξε ε, το θέμα της παραγράφου 6. Παράγραφος 17 Τροπολογία 238. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 17. Α, 239, συγγνώμη, παράγραφος 17. Καταπίπτει λόγω της 238. Προχωρούμε στη συμβιβαστική ε, C21. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 247. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 248 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 249 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω το 249 εγώ. Έχω 247, 248 και μετά πάει στο 250. 249 ο εισηγητής. Το 249 καλύφθηκε από τη συμβαστική 15. δεν το λέει αυτό στις σημειώσεις μου, λέει η πρόεδρος. Η πρόεδρος. Εάν συμφωνεί ο εισηγητής ότι έχει καλυφθεί το 249, εντάξει, ωραία. Τότε προχωράμε στη 250 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Καλύτερα όμως να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 250 παρακαλώ ψηφίστε. Πέρασε τη ψηφοφορίας, δεκτή. Παράγραφος 19, αρχικό κείμενο, υπέρ κατά αποχές δεκτό. 251 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 252 υπέρ κατά αποχές δεκτή, δεκτή 253 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 254 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αρχικό πρότυπο κείμενο της παραγράφου 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή δεκτό. Ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι έγινε δεκτή. Αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 3. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Δεκτή, δεκτή η τροπολογία 3. Σαφέστατα. Συμβιβαστική C1 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή αρχικό κείμενο ε, του, του εκτιμώντας β υπέρ κατά αποχές δεκτό ε, τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή υπέρ κατά αποχές δεκτή τώρα μια γλωσσική τροπολογία δεν χρειάζεται ψήφιση η 13 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική C2 υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, προχωρούμε στην 22 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι έγινε δεκτή. Α ελέγξουν ηλεκτρονικά τροπολογία 22, παρακαλώ. Ψηφίσατε. Έχουμε ένα παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Μία επιπλέον ψήφο. Τώρα είμαστε εντάξει, πέρα στις ψηφοφορίες Ωραία δεκτή. 27. Υπέρ, κατά, αποχές. έχει καταπίπτει 27 και 23. Ωραία, προχωράμε στην τροπολογία 30. Α, και αυτή καταπίπτει. 24. Υπέρ, κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική C4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική C5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Α, είναι το πρώτο τμήμα. Αυτό ήταν το πρώτο τμήμα, λέει η πρόεδρο. Το δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ το δεύτερο τμήμα. C5. Ψηφίσατε. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προχωρούμε στην τροπολογία 37. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι έγινε δεκτή. Παρακαλώ, ηλεκτρονική ψηφοφορία 37. Ψηφίσατε. Δεκτή. Αλλά με μικρή διαφορά. Τροπολογία 40. Ως προσθήκη. Τροπολογία 40. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συνεβαστική 6. C6 που έχει ένα νέο τμήμα στο μέσον στο οποίο έχουν συμφωνήσει όλοι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή προχωράμε στην συμβαστική C7 και πάλι ε, αναφέρεται στο detail transaction λεπτομερείς συναλλαγές υπέρ κατά αποχές δεκτή προχωρούμε τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προχωρούμε στην συμβαστική 23. Ο κύριος Κάμπεν Μετά τη χτεσινή συζήτηση που έγινε για αυτό το θέμα και για τη διάρθρωση του και ή διαζευτικού ή, ε, προτείναμε μια προσπάθεια γλωσσικού συμβιβασμού που να λέει και λέω στα αγγλικά τρίτη γραμμή και ε, ευρωπαϊκό νόμισμα και ευρωπαϊκή οντότητα ή σχετικά με ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ευρήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο λύσεις που δεν μας κάνουν, γιατί στη μία περίπτωση είναι πολύ ευρύ το θέμα και χρειάζονται και τρεις προϋποθέσεις ή στην άλλη περίπτωση μία από τις μία προϋποθέσεις μόνον υπάρχει που ούτε και αυτό μας κάνει και γι' αυτό λέμε η πρώτη προϋπόθεση να είναι υποχρεωτική με τη δεύτερη ή η πρώτη με την τρίτη. Οπότε είναι ένα συν δύο ή ένα συν τρία νομίζω ότι γλωσσικά ξεκαθαρίζεται κάπως το πράγμα και είναι πιο κατανοητό σε όλες τις γλώσσες, γιατί όντω υπάρχουν προβλήματα στις διάφορες γλώσσες με το κόμμα, δηλαδή όταν βάλουμε και ε, συμπληρώνεται αυτό το και με ένα μέρος, το επόμενο ή όχι. Οπότε ευρωπαϊκό νόμισμα και το δεύτερο ή το πρώτο με το τρίτο. Μάλιστα. Είχαμε αυτή τη συζήτηση εχθές και είχαμε πει ότι θα κάνουμε ε, ε, ψηφοφορία, το ότι να, τώρα έχω αντίρρηση να έρθει αυτή η πρόταση την τελευταία στιγμή. Η πρόεδρος, δεν είμαι βέβαιη ότι με αυτό που προτείνετε εσείς θα λειτουργήσει το, ε, το, το, το ουσιαστικό περιεχόμενο ε, μπορούμε βεβαίως να το οριστικοποιήσουμε στην Ολομέλεια, αλλά αυτό που προτείνω τώρα να κάνουμε είναι να την ψηφίσουμε όπως είχε προταθεί αρχικά. Ο εισηγητής, ο κύριος Λάγκε, προτείνω να ψηφίσουμε και μετά έχουμε τη δυνατότητα διόρθωσης καθοδών προς την Ολομέλεια. Το, εάν χρησιμοποιήσουμε το και, οι προϋποθέσεις είναι τρεις. Εάν χρησιμοποιήσουμε το διαζευτικό ή, τότε έχουμε δύο από τις τρεις ε, εναλλακτικές λύσεις. Εχτες είπαμε, πιστεύω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν να αφήσουμε το και και στα δύο σημεία. Να μείνει το και και στα δύο σημεία. Εντάξει λέει πρόεδρος, τότε ψηφίζουμε τροπολογία 23 στην αρχική της μορφή, υπέρ. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Δεν, δεν ακούμε. Η πρόεδρος λέει ότι η προφορική τροπολογία κατέπεσε διότι υπήρξε αντίρρηση διαδικαστική. Δεν ισχύει. Υπάρχει τυπική επίσημη αντίρρηση στην προφορική τροπολογία που παρουσιάστηκε μόλις τώρα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Ο εισηγητής προτείνει να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο το οποίο το είχαμε χτες αλλά δεν νομίζω να υπάρχει πλειοψηφία επ' αυτού. Εγώ ήθελα να καταλάβω αν η αντίρρηση του εισηγητή ήταν μόνο στην πρόταση προφορικής τροπολογίας του κυρίου Καμφέν ή αν αναφερόταν και στην προφορική τροπολογία που έχει υποβάλει η δική μου ομάδα. Ε, λοιπόν, πρόκειται για το εξή λέω εισηγητή. Το συζητήσαμε επισταμένως εχθές. Η ομάδα μου είναι το, το μόνο σημείο που μου ζήτησε η ομάδα μου ότι δεν πρέπει να υποχωρήσω και να παραμείνουμε στο και. Εάν θέλετε μπορούμε να ψηφίσουμε το και ή το ή. Το αποτέλεσμα θα φανεί. Το επίσημη αντίρρηση όμως έχει καταγραφεί. Η πρόεδρος, η προφορική τροπολογία είναι σε δύο τμήματα. Αυτό που θα κάνουμε είναι, θα ψηφίσουμε την συμβιβαστική 23. Μετά θα ψηφίσουμε την αρχική διατύπωση που λέει and to which an EU financial institution και στο οποίο ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κλπ. Με το end. Θα δούμε αν υπά... πού υπάρχει πλειοψηφία. Ας ψηφίσουμε καταρχάς τη συμβιβαστική 23 με το και. Με το end υπέρ. Κατά, αποχές ε, δεκτή κύριε Μπούλμαν δεκτή δεκτή και χωρίς την ομάδα σας έτσι κι έγινε δεκτή υπερψηφίστηκε κυρία Πρόεδρε κοιτάξτε εδώ δεν, κάνουμε, δεν παλεύουμε μεταξύ μας. Υπάρχει ο κανονισμός ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λογική λύση σε περίπλοκα προβλήματα. Η ομάδα μου έχει την εξής θέση. Ότι για οι τροπολογίες οι μας του κύριου Ντομίνιτσι αυτές τις υπερψηφίζουμε. Επίσης θα υπερψηφίζαμε την προφορική τροπολογία αν ήταν δυνατόν όμως θα ψηφίζαμε και για το πνεύμα του εισηγητή, για την αρχική διατύπωση, αν είχαν υπορριφθεί οι άλλες δύο περιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να εκφραστούμε. Ανατρέψτε λοιπόν τη σειρά. Εάν ψηφίσουμε τώρα την συμβιβαστική 23 ως έχει, δεν μπορούμε να την υπερψηφίσουμε. Πρέπει να την καταψηφίσουμε. Η Πρόεδρος. Εάν θέλετε να ψηφίσουμε το και ή το ή, τότε μπορώ να το δεχθώ. Όμως την περασμένη φορά που το πρότεινα είχατε αντιρρήσεις να ψηφίσουμε με αυτή τη σειρά. Ίσως τώρα είδατε ότι αυτή η λύση είναι η πιο λογική. Πιστεύω ότι πρέπει πάντοτε να ψηφίζουμε πρώτα τα, τις μίνι τροπολογίες και μετά τις μεγάλες τροπολογίες. Ο κύριος Μπούλμαν, κοιτάξτε, ποιος, ποιος, ποιος έχει κερδίσει τώρα από όλη αυτή τη ε, συζήτηση που έχουμε κάνει εδώ. Μάλλον σύγχυση επικρατεί. Η πρόεδρος. Εγώ νομίζω ότι τελικά μου δώσατε δίκαιο με αυτά που είχα προτείνει εχθές. Θα ψηφίσουμε, λέει η πρόεδρος, το και έναντι του διαζευτικού «η». Υπέρ. Το «ε». Το «end». «End», λέει η πρόεδρος. Υπέρ και όσοι θέλουν το «ή», το διαζευτικό. Ποιος κέρδισε. Το «ΕΝΤ». Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Παρακαλώ ψηφίστε όσοι είναι υπέρ του «και». Ψηφίσατε όλοι. Τρεις ψήφοι λείπουν ακόμα. Παρακαλώ ψηφίστε όλοι. Έληξε η ψηφοφορία. Κέρδισε το and, το και. Άρα καταπίπτει το or, το e. Επιστρέφουμε τώρα στην, ψηφοφορία τη συμβαστική 23 με το END και έγινε δεκτή, υπέρ κατά δεκτή. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει προηγούμενο μέσο συμφωνίας. Πρώτα ψηφίζουμε τα μήνυ, τα μικρά, τα εσωτερικά και μετά ολόκληρη τροπολογία. Λοιπόν, 73 υπέρ κατά αποχές 73. Παρακαλώ, απορρίπτεται λέει η πρόεδρος. δεν ήταν σαφές τι, τι, ψήφισε το ΕΛΚ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, παρακαλώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 3, 3 της ΔΕΒΕ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε τώρα το κείμενο ως τροποποιηθέν. Παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία του κειμένου έτσι όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίσατε πέρα τις ψηφοφορίες, 43, 43 ψήφοι υπέρ, μία κατά συγχαρητήρια στον κύριο Λάγκα. Τώρα. Εντάξει. Ίσως τώρα μπορούμε να επιταχύνουμε κάπως. Εδώ έχουμε την ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης ε, του κυρίου Σικλούνα για την υιοθέτηση από πλευράς Εστονίας του ενιαίου νομίσματος. Ναι, ξέρω έχετε όλοι εδώ τώρα ενθουσιαστεί με αυτή την ψηφοφορία αλλά είναι και αυτό εδώ πολύ σπουδαίο ότι έχουμε ένα κράτος μέλος που πιστεύει ότι πιθανότατα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις για να μπει στο ευρώ. Μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνη στο ευρώ. Uh, Ψήφι τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, τροπο, ε, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 9 του πρωτότυπου κειμένου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφοι 11 με 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Εκτιμώντας α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο εκτιμώντας β και γ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται και οι αναφορές unblock, η αιτιολογική σκέψη unblock υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τελική ψηφοφορία για το κείμενο. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, ευχαριστώ. Πέρασε τη ψηφοφορία. 40 υπέρ, 2 κατά, μια αποχή, εγκρίνεται. So, congratulations to the rapporteur. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και συγχαρητήρια στην Εστονία. Right. We now move on. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης του Χαρίτερ Μάρτιν για την σύνδεση των μητρών των επιχειρήσεων. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τα μηνύματα που στέλνετε. Να το ελέγξουμε. Has everybody voted? Okay, votes closed. Ψηφίσατε όλοι, απορρίπτεται. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 3. Α, ναι, συγγνώμη. Πρέπει να ψηφίσουμε για το πρωτότυπο κείμενο. Της παραγράφου 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε την τροπολογία 4 παρακαλώ ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται Πρώτο κείμενο παράγραφος 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4 πρώτο κείμενο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική για την παράγραφο 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική β υπέρ. Κατά αποχές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 Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το κείμενο που τροποποιήθηκε. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Okay, we Περνάμε τώρα στην εξέταση του σχεδίου έκθεσης του Ότμαρ Κάρας. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση της ε, οδηγίας για τα CRD4, δηλαδή για τις ε, απαιτήσεις κεφαλαίου. tariffs. Right, I think it's uh, quiet enough now. Right. Mr. Karas, the floor is yours. Κύριε Κάρας, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Ε, θέλω να παρουσιάσω σύντομα το σχέδιο γνωμοδότησης. Τι, έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά τα θέματα και έχουμε πει ακριβώς γιατί χρειαζόμαστε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Κατά την άποψή μου αυτή η έκθεση γίνεται όλο και πιο σημαντική από μέρα σε μέρα και δει συζήτηση στην Επιτροπή μας. Γιατί? Διότι η εισηγήτρια του CAD3 είναι εδώ και οι Αμερικανοί μας λένε ότι δεν σε εφαρμόσουν όλα τα σημεία του CAD3. Στο 2 είχαν την εμπειρία ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν υλοποίησαν, δεν εφάρμοσαν τη Βασιλεία 2. Άσχετα λοιπόν από αυτή την εμπειρία, αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή της Βασιλείας, όπως τη λέμε CAD 4 ή Βασιλεία 3, συζητείται έντονα και το πρόγραμμα είναι να ολοκληρωθεί και να ψηφιστεί μετά το καλοκαίρι. Και η Κομισιόν μας υπέβαλε ε, ένα σχέδιο οδηγίας επί της Βασιλείας ε, και γι' αυτό πρέπει ακριβώς να παρέμβουμε και να συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν το περιεχόμενο αλλά και τη θέση ενισχύ πότε ακριβώς θα τεθεί σε εφαρμογή και τα συναφή θέματα. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να αναλάβει έναν υπεύθυνο ρόλο και να μας αναφέρει τι συμβαίνει, τι γίνεται στην Επιτροπή Βασιλεία και να συντονίσει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση, το είδαμε και στην ακρόασή μας, δεν δημιουργεί ένα σεμιτό επίπεδο για τους κανόνες του παιχνιδιού και υπάρχει μεγάλη διαφορά στο πώς ενεργούν οι τράπεζες και πώς καθορίζουν, πώς ορίζουν το, την ποιότητα του κεφαλαίου και τι χρειάζεται, τι μέτρα πρέπει να εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφορά μεταξύ πραγματικότητας και θεωρητικών συζητήσεων στην Επιτροπή της Βασιλείας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία ενδελεχή ανάλυση από πλευράς Κομισιόν διότι μία μελέτη για τις τράπεζες δεν αρκεί. Βεβαίως έχουμε δεσμευτεί έναντι του στόχου των G20 για την ποιότητα του κεφαλαίου και ότι πρέπει να ενισχυθεί η ποιότητα του κεφαλαίου και να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο. Πρέπει όμως να βρούμε μια καλή ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων, ε, νομοθετικών ρυθμίσεων και χρηματοδοτικών πόρων. Διαθροτικές ανισορροπίες και η, ανισορροπία που υπάρχει στην παρούσα πρόταση δεν διασφαλίζουν την ανάκαμψη και μάλλον θα ζημιώσουν την ε, οικονομία της Ευρώπης. Πρέπει να είναι αποφασιστικές οι συνθήκες ανταγωνισμού διεθνώς. Αυτή τη στιγμή η Αμερική δεν είναι πρόθυμοι, δεν θέλουν να προσαρμόσουν τους κανόνες των ισολογισμών με τις διατάξεις περί ανάληψης κινδύνου. Θέλουν το ρίσκο ε, να αναφέρεται, να ενταχθεί στα στοιχεία του ισολογισμού μόνο όταν έχει πλέον φτάσει σε επικίνδυνη κατάσταση. Ενώ εμείς θέλουμε μία διαρκή αξιολόγηση του κινδύνου από το α μέχρι το ω. Δεδομένου ότι ο κίνδυνος αυτός έχει επίπτωση στα κεφάλαια και στην κεφαλογική δομή. Εάν λοιπόν δεν συμβεί το ίδιο, εάν δεν εφαρμοστούν ίδια μέτρα από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, δεν θα επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Τώρα, για την ποιότητα του κεφαλαίου εμείς έχουμε μία οικονομία η οποία κατά, τις, ο, κατά 80% ε, κινείται μέσω δανείων. Χρηματοδοτείται από δάνεια, από συνεταιριστικές τράπεζες, εμπορικές τράπεζες, ε, ιδιωτικές τράπεζες. Έχουμε λοιπόν μία διαφορετικές δομές οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη έναντι των της άλλης πλευράς του Ατλαντικού και πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, του, των χρηματιστηρίων και των χρηματοδοτικών εργαλείων. Δεν θέλουμε να μειώσουμε τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών, αλλά θέλουμε να αυξήσουμε την ποιότητά τους. Όσον αφορά τώρα τα, τα πρότυπα Θέλουμε να αναπτύξουμε ρευστότητα υψηλής ποιότητας και ε, να μειώσουμε τον κίνδυνο να μαζευτεί ρευστότητα σε ένα υπερβολική ρευστότητα σε ένα σημείο ενώ αλλού να μην υπάρχει καθόλου ρευστότητα και να υπάρχει τεράστια στενότητα όσον αφορά την παροχή δανείων. Θέλουμε επίσης να εφαρμόσουμε ένα δίκτυ μόχλευσης ε, σαν ένα πιθανό ανάχωμα, μια πιθανή προστασία έναντι της υπερβολικής μόχλευσης. Το, ο ΔΕΛΤΑ ο δείκτης μόχλευσης, ε, κινδυνεύει να θίξει την Ευρώπη πολύ αρνητικά όταν σε άλλες περιφέρειες, σε άλλες περιοχές της γης ο δείκτης μόχλευσης χρησιμοποιείται πολύ πιο ευέλικτα για την ε, χρηματοδότηση. Οι, στρατη... οι τραπεζικές στρατηγικές πρέπει να διαφοροποιούνται. Το one size fits all, δηλαδή ε, ένα μοντέλο ε, ταιριάζει σε όλους, δεν είναι σωστό, δεν λειτουργεί σωστά. Πρέπει να διαφοροποιηθούμε και να υπάρχουν και βασμοί ευελιξίας όλες οι νομοθετικές προτάσεις για, για τις τράπεζες πρέπει να είναι συνεκτικές. Να υπάρχει μία συνοχή. Και η, στα συμπεράσματα πρέπει να αξιολογήσουμε όλες τις προτάσεις και σας ε, ζητώ, κάνω μία έντονη έκκληση να θεωρηθούμε όλοι υπεύθυνοι για το τελικό αποτέλεσμα της Βασιλείας και να μην το αφήσουμε το θέμα αυτό τελείως στα χέρια της Κομισιόν και της ε, αναθεωρημένης ε, οδηγίας, διότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, γιατί η Βασιλεία 2 είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία της Ευρώπης και για τις αγορές. Έχουμε ακόμα καιρό να επηρεάσουμε τα πράγματα. Ζητώ από την Επιτροπή της Βασιλείας να συζητήσει τα θέματα αυτά τα οποία αναφέρω εγώ στο σχέδιο γνωμιδότησης και να τα συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των διαβολεύσεων το, κατά την καλοκαιρινή και την περίοδο και τη φθινοπορεινή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι ο κ. Λούλινγκ πρέπει να φύγει και κανονικά θα έπρεπε πρώτα το σκιώδης, αλλά εφόσον ο κ. Λούλινγκ πρέπει να φύγει, Εντάξει, θα της δώσω το λόγο μετά όμως από τον Ρούντολφ. Ευχαριστώ, λέει ο Ούντο. Τρία βασικά σημεία από τη δική μας πλευρά. Πιστεύουμε ότι τα κεφάλαια θα πρέπει να είναι ε, ε, δεν εμπλουτιστούν, να έχουν καλύτερη ποιότητα, αλλά πρέπει να είμαστε έξυπνοι στο πώς θα χειριστούμε το θέμα των κεφαλαίων, διότι εάν δεν καταφέρουμε μια σωστή διαχείριση και μια προσφορά σωστών ποιοτικών κεφαλαίων, θα αποτύχουμε. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά. Όπως είπε και ο συγγήτης, δεύτερον, κάθε χρηματοοικονομική αγορά έχει το δικαίωμα να ε, διασφαλίζει τα, τα ίδια της κεφάλαια. Τώρα όλοι θέλουν να αναθεωρήσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές, όλοι θέλουν να εξασφαλίσουν μια βελτιωμένη ποιότητα των κεφαλαίων τους, αλλά πολλές φορές πιεζόμε, πιεζόμαστε από την διεθνή ανταγωνιστική πολιτική. Μας πιέζει ο ανταγωνισμός. Οι συνθήκες των συναλλαγών επηρεάζονται από συγκεκριμένες προτάσεις, ρυθμιστικές προτάσεις. Πρέπει λοιπόν να προβάλλουμε, να αποφασίσουμε συγκεκριμένες ε, ρυθμιστικές, συγκεκριμένους ρυθμιστικούς κανόνες για να μπορούν να λειτουργήσουν οι αγορές σωστά. Ε, το, ευρωπαϊκό, το, το τραπεζικό σύστημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο και πώς θα προχωρήσουμε με το δίκτυ μόχλευσης ο δίκτυς μόχλευσης πρέπει να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, λογικούς περιορισμούς όσον αφορά τους κινδύνους. Δεν πρέπει να καθορίσουμε εδώ ε, τυχαία ποσοστά ή τυχαία τυχαίους αριθμούς για τον περιορισμό του δίκτυα αλλά πρέπει να προσαρμόζεται, να, είναι, να έχει μία ευελιξία όσον αφορά το ύψος του κινδύνου και όχι έτσι να καθορίσουμε αυθαίρετα μια συγκεκριμένη αξία του δίκτυ. Χρειαζόμαστε λοιπόν πλήρη ανάλυση που να μας λέει τι πρέπει να ρυθμιστεί και τι δεν πρέπει να ρυθμιστεί. Και επίσης να γνωρίζουμε ακριβώς ε, ποιο είναι το υπόβαθρο των προτάσεων που προέρχονται από την Επιτροπή της Βασιλείας και την Κομισιόν. Εμείς δεν θα δεχτούμε εν ώψη της κρίσης φορείς οι οποίοι αυτορυθμίζονται να προσπαθήσουν να μας αντικαταστήσουν ως νομοθέτες. Δεν είναι δυνατόν αυτορυθμιζόμενοι φορείς όπως η Επιτροπή της Βασιλείας να αντικαταστήσουν δημοκρατικά εκλεγμένους φορείς και αυθαίρετα να αποφασίσουν κανόνες και ρυθμίσεις που αντιτίθενται στις, ε, στη λογική ή στις, ε, στο, διεθνή ανταγωνισμό. Γι' αυτό, όπως είπε και ο συγητής, έχουμε ακόμα περιθώριο να παρέμβουμε στη διαδικασία της Επιτροπής της Βασιλείας και να ζητήσουμε ε, μία πλήρη ανάλυση των προθέσεων τους. Πιστεύω ότι το σχέδιο γνωμοδότησης του έτσι όπως έχει σήμερα είναι πολύ καλό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ε, Σκιώδης Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικές παρατηρήσεις. Το πρώτο σχέδιο αυτογνωμοδότησης ε, έχει πολλά θετικά σημεία. Συμφωνώ βασικά με τον Ούντο ότι πρέπει να επιτύχουμε μια ευρεία συνένεση. Μερικές παρατηρήσεις. Πρώτον, για τα πρότυπα ρευστότητα. Οι κανόνες για τα πρότυπα ρευστότητα που προτείνονται από την Κομισιόν δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν, δεν θα εφαρμόζονται σε επενδυτικές εταιρείες εκ μέρους των πελατών τους. Εδώ ακριβώς υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Τι κάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για δικό τους συμφέρον και τι κάνουν για το συμφέρον των πελατών τους. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια εδώ, διότι δεν θέλουμε να ανοίξουν παραθυράκια που να παρακάμπτουν την νομοθεσία. Δεύτερον, ο ορισμός του, του, κεφαλαίου. Εδώ πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα πάρα πολύ απλά και με κεφάλαιο να εννοούμε ε, με, μετοχικό κεφάλαιο και πόροι και resources, πόροι για την λευστότητα και τον δίκτυ, δίκτυ μόχλευσης ο δείκτης μόχλευσης έχουμε εδώ έναν ορισμό αλλά δεν έχουμε καμία αναφορά στον περιορισμό ε, του δείκτη αυτού. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε ότι υπάρχει ε, η απόλυτη ανάγκη να υπάρχει μία οροφή, μία οροφή της μόχλευσης και πιστεύω ότι η έκθεση πρέπει να τροποποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση η μόχλευση είναι αυτά τα οποία δεν βρίσκονται, δεν υπάρχουν στον ισολογισμό. Οπότε πιστεύουμε, αντί να προσπαθήσουμε μέσα στο δίκτυ μόχλευσης να καλύψουμε όλα τα οποία είναι off-balance sheet, εκτός ισολογισμού, να ενεργήσουμε αντίθετα και να προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε τα πάντα στον ισολογισμό ό,τι είναι off-balance sheet, πολλές φορές οι τράπεζες ξεφεύγουν από τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό ακριβώς τα βγάζουν από τον ισολογισμό. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε από τις τράπεζες τι βρίσκεται εκτός ισολογισμού. Πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε τα εκτός ισολογισμού στοιχεία στα, στο μίνιμουμ, στο ελάχιστο, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια με τα στοιχεία που αναφέρονται στους ισολογισμούς. Και τέλος, τα αντικυκλικά μέτρα το μεγάλο πρόβλημα που βλέπουμε είναι η αξιολόγηση του κινδύνου. Η αξιολόγηση του κινδύνου γίνεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα ίδια και έχουν ε, ακριβώς πολλά προηγούμενα, έχουμε πάρα πολλά προηγούμενα ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είτε δεν θέλουν είτε δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν σωστά τον κίνδυνο. Άρα λοιπόν ε, πολλές φορές καταφεύγουν σε εξωτερικούς ε, συμβούλους ή σε εξωτερικούς φορείς αξιολόγησης του κινδύνου και έτσι δημιουργείται μια ολόκληρη καινούρια ιστορία, μια νέα επιχείρηση. Σε ορισμένους αρέσει αυτή η προσφυγή σε τρίτους. μια νεα επιχειρηση σε αρεσει αυτη η προσφυγη σε τριτους αλλα τα, τα θέματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Εγώ πιστεύω ότι, ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι διατάξεις που να τους υποχρεώνουν σε, έναν αντικειμενική, σε μια αντικειμενική αξιολόγηση κινδύνου και όχι αξιολόγηση του κινδύνου να γίνεται έτσι όπως τους συμφέρει. Ο στόχος μας πρέπει να είναι απλούστευση, απλές διαδικασίες, όχι περιπλοκότητα, διότι η περιπλοκότητα ανοίγει την πόρτα στους κινδύνου. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε την, ε, τις απλές, ε, τους απλούς κανονισμούς ότι θέλουμε να διέπονται από μια προσέγγιση απλότητος, δηλαδή διαφάνειας και σαφήνειας. Ένα θέμα που δεν είδαμε να αναφέρεται στο σχέδιο γνωμοδότησης είναι ότι θα πρέπει αναλογικά με το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να αυξάνεται και το μέγεθος των κεφαλαίων. Να υπάρχει δηλαδή μια σταδιακή αύξηση των κεφαλαίων εφόσον αυξάνεται το μέγεθος του ιδρύματος. Ε, ε, τώρα επανέρχομαι στην προσέγγιση του narrow banking, της στενής ε, τραπεζικής δραστηριότητας ξέρω για ορισμένους από εσά οι ρυθμίσεις αυτές ε, που προτείνονται είναι υπερβολικά σκληρές και όχι βιώσιμες. Αυτό που μπορούμε να προτείνουμε είναι να μειώσουμε τις κεφαλουχικές απαιτήσει των τραπεζών όταν οι τράπεζες μειώνουν το εύρος των δραστηριοτήτων τους. Δηλαδή, εάν μια τράπεζα από ε, τεράστια θέλει να γίνει μικρότερη, να, περιορίσει δηλαδή τις δραστηριότητες της και να ονομαστεί narrow, να κάνει narrow banking, τότε μπορούμε ίσως να ζητήσουμε ε, λιγότερο αυστηρές διατάξεις για τα κεφάλαιά τους, για την, ε, ε, τα αναγκαστικά αποθέματα κεφαλαίου που πρέπει να έχουν. Ίσως όταν μια τράπεζα λοιπόν, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μετακινείται προς το στενό μοντέλο λειτουργίας μπορούμε να στενέψουμε και τις απαιτήσεις των κεφαλουχικών τους αποθεμάτων. Ευχαριστώ. Βίκη, εσύ είσαι σκιώδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότμαρ, για την εξαιρετική σου έκθεση, που νομίζω ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ και έχει μιλάει για περίπλοκα πράγματα με πιο ευκολονόητο τρόπο. Πιστεύω πως αυτή είναι πολύ έξυπνη προσέγγιση. Είναι περίπλοκη ε, και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας καθοδηγήσεις. Σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σου. Ε, όντως ε, χρειάζεται να συντονιστεί το χρονοδιάγραμμα αλλά και να συντονιστούμε με τους είπα και να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπούλμαν για τη διαφάνεια σχέσης με τη Βασιλεία που μίλησε. Είχαμε μια πολύ καλή διάσκεψη με το CRD3 με τη Βασιλεία και ότι είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπουμε τον αντίκτυπο να ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους άμεσα. Ε, δηλαδή να βλέπουμε ποιος είναι ο αντίκτυπος των όσων νομοθετούμε εδώ. Ευχαριστώ επίσης για τα όσα είπες για την ε, ανάγκη να εστιάσουμε στη διεθνή λογιστικά πρότυπα. Γιατί εφόσον θέλουμε διεθνή νομοθεσία θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε και το θέμα των διεθνών λογιστικών σταντάρ. και δεν αρκούν κάποιες, ε, κάποιες χώρες να λένε ότι εγώ θέλω διαφορετικά να ρυθμίζω κάποια πράγματα. Τώρα, για το θέμα που αναφέρθηκε και στην τελευταία συζήτηση, ε, θα πρέπει όντω να δούμε τι είναι μια ρευστή αξία. Μπορεί δηλαδή οι τράπεζες να κατέχουν χρέη κρατών ως ε, ρευστή αξία και τα κράτη μετά να δυσκολεύονται. Είναι πολύ σημαντικό και λεπτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, εάν συμπεριλάβουμε για παράδειγμα τα, τα ομόλογα κάλυψη, εκεί μπορεί να οδηγηθούμε σε συστημικά προβλήματα όσον αφορά την αγορά. Θα πρέπει λοιπόν πολύ σοβαρά να σκεφτούμε τι συμπεριλαμβάνει η ρευστότητα. Για τον ορισμό του κεφαλαίου, άκουσα τα όσα είπατε για το ότι θέλετε να έχουμε το κεφάλαιο όσο γίνεται πιο ξεκάθαρο, γιατί το κεφάλαιο πρέπει να καλύπτει τις απώλειες πριν μια τράπεζα χρεοκοπήσει. Ωστόσο υπάρχουν διάφορα θέματα. Έχουμε διάφορους ομίλους επιχειρήσεων, ας πούμε στη δικιά μου χώρα, που δεν ε, είναι εγγεγραμμένοι στο χρηματιστήριο και, και οι οποίες είναι ιδιοκτησία των ίδιων τους των πελατών. Και αυτό ήταν ένας πολύ σταθερός τρόπος για την εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα τους επηρεάσουμε αυτού αρνητικά. Τώρα, ε, για τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν οι τράπεζες στην ευρύτερη οικονομία είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Ήμουν και εγώ ε, μέλος και γνωρίζω πολύ καλά το τι έκαναν οι τράπεζες για την κατασκευή των υποδομών, των τηλεπικοινωνιών, ε, του δικτύου του ενεργειακού και πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Το 2020 έχουμε την ψηφιακή ημερήσια διάταξη, πρέπει να εξετάσουμε διαφορετικά την ενέργειά μας και όλα αυτά χρειάζονται κεφάλαια. Είναι πολύ σημαντικό οι τράπεζε λοιπόν να συνεχίσουν να παίζουν ε, τον ρόλο τη παροχή των χρημάτων για την υλοποίηση αυτών των ε, σχεδίων. Το θέμα είναι να δούμε πόσο εξαρτάται η Ένωση από την χρηματοδότηση των τραπεζών σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου. Όταν ορίζουμε λοιπόν τι κάνουν οι τράπεζε, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις άλλε λειτουργίε που δεν είναι μόνο ο δανεισμό. και ο ένας από του ρόλου είναι η σύνδεση που παίζουν οι ρόλοι, ο συνδετικό ρόλο που παίζουν οι τράπεζε. ανάμεσα μέσα σε αυτούς που χρειάζονται τις επενδύσεις και αυτούς που επενδύουν, τους επενδυτές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός ε, τομέας. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς ε, όντως ε, η τιτλοποίηση προχώρησε τόσο πολύ, αλλά ε, αυτή τη φορά να φτάσουμε σε μια σωστή ισορροπία. Συμφωνώ και με διάφορα άλλα πράγματα. Θα πρέπει να σκεφτούμε και διάφορα άλλα που έχουν κάνει οι τράπεζες για την παγίωση των οικονομικών αγορών. Έχουν βοηθήσει τις εταιρείες να αναλάβουν τέτοιους κινδύνους. Γι' αυτό και θα πρέπει να διευρύνουμε κάπως την έννοια του τι αξίζει, τι προσφέρουν οι τράπεζες στην κοινωνία μας και όταν θα εξετάζουμε παράλληλα τον αντίκτυπο που θα έχουν όλα αυτά στο τραπεζικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Άστριτ, θέλεις τώρα να παρεμβείς, γιατί νομίζω ότι μετά πρέπει να φύγεις. Ευχαριστώ. Πρέπει να ασχοληθώ με το βιολογικό κρασί στην Επιτροπή Γεωργίας μετά. Γι' αυτό και... Καταλαβαίνετε, είναι σημαντικό, ε? Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να φύγω. Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ εδώ να στηρίξω λίγο τη γενική γραμμή του εισηγητή μας. Το ξέρει εξάλλου ότι βρίσκω καλά αυτά που μας λέει. Πραγματικά έχει μια σωστή αντιμετώπιση. Η οδηγία λοιπόν αποσυνδέει τους ίδιους πόρους. Είναι μια οδηγία η οποία θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική στιγμή όσον αφορά το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Τις εξελίξεις θέλουμε να τις προετοιμάσουμε κάτω από τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες. Ιδιαίτερα μάλιστα γιατί θέλουμε να ανταποκριθούμε σε κάποιες απαιτήσει με αυστηρότητα γιατί είναι αναγκαίο εξαιτία της οικονομικής κρίσης. Όμως επιμένω και δεν, νομίζω, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και πολλοί συνάδελφοι μαζί μου, επιμένω για το ότι δεν πρέπει από την άλλη μεριά να πνίξουμε τον τομέα με περιορισμούς τόσο αυστηρούς που τελικά ολόκληρη η ευρωπαϊκή οικονομία να ζημιωθεί. Όντως είναι πραγματικά μια άσκηση ακροβατισμού και νομίζω ότι ο ρόλος του εισηγητή μας εδώ είναι δύσκολος. Πρέπει να εξετάζουμε τα πράγματα χωρίς ε, να έχουμε προκαταλήψεις, με μετριοπάθεια. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Συμφωνώ λοιπόν με τα περισσότερα τα οποία μας παρουσίασε ο εισηγητής. Θέλω όμως, επιτρέψτε μου, να εκφραστώ πάνω σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Το θέμα είναι το ένα, ο δείκτης μόχλευσης. Μας έχει δοθεί και άλλη φορά η ευκαιρία να συζητήσουμε γι' αυτό. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να τον δούμε σαν κάτι το ουδέτερο. Γιατί όταν έχει να κάνει με ασφαλή προϊόντα, εγκυμένα, τότε ο δείκτης μόχλευσης δεν παίζει κανένα ρόλο. Μόνο από τη στιγμή που έχει να κάνει με πιο επικίνδυνα προϊόντα, κερδοσκοπικά, τότε μόνο τίθεται το ζήτημα. Εξού και η ερώτησή μου που μπορεί να σας φανεί αφελής. Αντί να εισάγουμε ένα ή πολλά κλάσματα, αναλογίες δηλαδή για το δίχτυ που να είναι άκαμπτα, δεν θα ήταν προτιμότερο να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα στην ε, ταξινόμηση με πραγματικούς κινδύνους. Νομίζω ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Και τι αν μη τι άλλο πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Και όχι να βάλουμε ένα γενικό κανόνα ο οποίος θα μπορούσε να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι για τα ταμιευτήρια. Και εδώ περιορίζουμε τις προϋποθέσεις άσκησης για τα ιδρύματα αυτά και φοβάμαι ότι εδώ πάμε υπερβολικά μακριά όταν εμποδίζουμε την άσκηση αυτής της λειτουργίας που είναι πολύ σημαντική σε πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Ο τομέας, βλέπετε, έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες του, το ξέρετε. Δεν θα ήθελα να μπω στις λεπτομέρειες εδώ, αλλά πάντως η αναλογία κάλυψης ρευστότητας πρέπει να προσαρμόζεται στις διάφορες δραστηριότητες των ε, τραπεζών αυτών των ταμιευτηρίων. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επενδύσεις ή για cover bonds, υποθήκες. Θέλω λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές και να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποια μαθήματα από την κρίση αυτή. Να ρυθμίζουμε εκεί που πρέπει να ρυθμίζουμε. Προσοχή να μην πνίξουμε, όπως είπα και στην αρχή, τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, ο οποίος μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχει να αναλάβει δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Ζητάω από τον εισηγητή λοιπόν και τον παρακαλώ να λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις μου αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Εγώ είμαι σκιώδης από πλευράς των φιλελεύθερων. Οπότε θα ήθελα εγώ να παρέμβω τώρα και μετά ο Ζαπόλο Καζέ και η κυρία Τζουρί. Πολλά από αυτά που ήθελα να πω έχουν ήδη υποθεί. Δεν θα τα επαναλάβω λοιπόν. Όμως, έχουμε να κάνουμε εδώ με πολλά από αυτά που έχει προβλέψει η Βασιλεία για πολλές μεγάλες τράπεζες, όχι για μικρές τράπεζες. Και ακριβώς εδώ είναι το ζήτημα, ότι δεν έχει να κάνει ούτε καν με όλες τις χώρες. Πρέπει λοιπόν τις διαφορές αυτές να τις λάβουμε υπόψη μας. Κυρίως σε μερικές χώρες όπου έχουν διαφορετικές δομές, ενώ άλλες χώρες όπως η δικιά μου, ίσως θέλουν να ανατρέψουν τις δυνατότητες που υπάρχουν αλληλασφάλισης για παράδειγμα. Αν θέλουμε να καλύψουμε αυτά που λέει ο κύριος Λάμπερτ για το narrow banking, πιο μικρές δομές, πιο ουδέτερες δομές, τότε πρέπει να φροντίσουμε ότι δεν θα κάνουμε κάτι που θα έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε, αν μπορούμε όντω να κάνουμε κάτι που να ενθαρρύνει αυτές τις νέε δομέ δεν ξέρω. Σίγουρα πάντως πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα από την άλλη μεριά. Τώρα, το θέμα του κυριαρχού χρέου. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο μηδενικός κίνδυνος προϋποθέτει ότι θα υπάρχουν αγορές ρευστότητας και ότι με το ευρώ δεν μπορούμε να τυπώσουμε καινούριο χρήμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ονομαστικός κίνδυνος. Μπορεί να υπάρξει. Ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να τυπώσουμε χρήματα. Και αυτό φάνηκε ότι υπάρχει κίνδυνος πιστότητας. Το είδαμε με την ελληνική κατάσταση. Άρα λοιπόν πρέπει να ερευνήσει κανείς. Αν δεν ήταν ε, για την αγορά κυρίαρχο χρέος από πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα υπήρχε. Βρέχει πρόθεσμα, πάντως δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μακροπρόθεσμα όμως, αν κοιτάξουμε τα πράγματα, πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση στην ευρύτερη δομή των όσο κάνουμε για την εποπτεία στην Ευρωζώνη. Ο, το Συμβούλιο το Νέο Συστημικού Κινδύνου θα έπρεπε να το δει αυτό και να προβλέψει κάποια πράγματα στην οδηγία για τα τρεπάρτια κεφαλαίου για την ποιότητα κεφαλαίου. Δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια τώρα θα διορθώσει το πρόβλημα. Με την νέα οδηγία, την 4, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όμως. Την CRD4. Το έχω σκεφτεί ξανά και ξανά, αλλά τώρα δημοσιεύτηκε. Δεν είπα τίποτα νωρίτερα, ακριβώς επειδή δεν είχε δημοσιευθεί ακόμα. Έπειτα, ποιο θα είναι το κεφάλαιο, πώς θα έχει καλή ποιότητα το κεφάλαιο. Πρέπει αν μη τι άλλο να δούμε κατάματα το γεγονός ότι έχουμε βρεθεί σε δύσκολη θέση εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχε αξιολογηθεί σωστά το κεφάλαιο ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Έρχομαι τώρα στα λογιστικά πρότυπα το I το έχετε βάλει αυτό. Πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να υπάρχει σύγκληση για τα πρότυπα που ισχύουν για τους επενδυτές και εκείνα που ισχύουν για εποπτικούς λόγους. Να ξεπεράσουμε το πρόβλημα ότι οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν την αξία των επιχειρήσεων εφόσον πολιθούν και οι επόπτες πρέπει να ξέρουν ποια θα είναι η σταθερότητα μακροπρόθεσμα. Και δεν υπάρχει ένα νέο λογιστικό πρότυπο το οποίο να καλύπτει και τις δύο αυτές απαιτήσει. Δεν θέλουμε να έχουμε δύο παράλληλους δρόμους, δύο παράλληλα πρότυπα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εφαρμόσουν την αρχή που λέει ότι το κάνετε για τους ε, επενδυτές, ετοιμάζετε τα πρότυπα και μετά βάζετε και κάτι για τη συνέχεια. Ορισμένοι έχουν διαμαρτυρηθεί. Γιατί τελικά αυτά απομακρύνονται από τα λογιστικά πρότυπα. Αλλά πρέπει να βρούμε μια στην πράξη ικανοποιητική λύση. Δεν θέλετε μια διτή γραμμή αναφοράς. Οι εκθέσεις δεν πρέπει να είναι παράλληλες, δεν μπορείτε να έχετε διαφορετικές αξίες για τους επενδυτές και άλλα αποτελέσματα για τον έλεγχο όχι. Άμα υπάρχει διαφάνεια και όλοι γνωρίζουν πώς το ένα νούμερο για τους επενδυτές γίνεται άλλο για τις απαιτήσει εποπτείας, είναι εντάξει ή όχι. Έρχομαι τώρα στην παράγραφό σας 13, όπου θέλετε να ενθαρρύνετε τις τράπεζες να βάζουν να διατηρούν τα δάνεια στα δικά τους βιβλία χωρίς υπερβολική τιτλοποίηση. Ε, ομόλογα δηλαδή. Γιατί αν θέλετε να είναι στα βιβλία τους, θα εφαρμόσετε και σε άλλα μέσα αυτό. Και η, τα καλυμμένα ομόλογα πολύ καλά για την εγκυμένα από τις τράπεζες. Αλλά οτιδήποτε καλύπτεται από τιτλοποίηση θα γίνεται τελικά καλυμμένο ομόλογα. Όπως στη Βασιλεία 2. Τότε όμως πρέπει να το δείτε και όσον αφορά την ευρύτερη έκθεση. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να έχετε τον δανεισμό που θέλετε αν δεν έχετε και ένα μηχανισμό για τις τράπεζες που να μπορούν να βγάλουν από τον ισολογισμό τους με υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο κάτι. Κάθε φορά που ελευθερώνεται κάτι που βγαίνει κάτι από τον ισολογισμό, από τα βιβλία τους, μετά πρέπει να μπορέσετε να συντεριάξετε τα κεφάλαια με αυτά που πάνε στην οικονομία. Ο δανεισμό λοιπόν βγαίνει από την πραγματική οικονομία μερικέ φορέ με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, στην παράγραφο 16 μιλάτε για του συνεταιρισμού και τα ταμιευτήρια. Εδώ ίσως θα πρέπει να βάλουμε και τα mutuals. Θα έπρεπε και αυτά να προσθεθούν πιστεύω γιατί είναι το γενικό ήθος που πρέπει να επικρατεί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και τέλος, όταν ερχόμαστε στον πιστοτικό κίνδυνο αντισυμβαλόμενων, να δούμε και αυτά που λέει έκθεση Λάγκεν. Και για τη μόχλευση, αυτό που είπατε κι εσείς θέλω κι εγώ να τονίσω. Να μην έχουμε στραβακίνητρα τελικά που εμφανίζονται. γιατί τότε επηρεάζεται όλο αυτό το θέμα του τι μπαίνει εκτός βιβλίων, τιτλοποίηση ή κάτι αντίστοιχο. Πρέπει όλα αυτά να γίνονται με υπεύθυνο τρόπο, ώστε να μπορεί κανείς να δανείζει στην πραγματική οικονομία. Και όχι απλώς επειδή φτάνει σε ένα όριο αυθαίρετο. Αυτά είναι τα σχόλια που είχα να κάνω εγώ. Και τώρα έχουμε άλλους τρεις. Τσούρι, Ζανπόλ Κοζές και Σερέρα. Α, ανάποδα. Όχι. Πρώτα είναι ο Ζαμπόλ Κοζές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάω εκ μέρους του ΕΛΚ. Εννοείται λοιπόν ότι στηρίζουμε απόλυτα τη δουλειά του συναδέρφου μας Κάρας και τη θέλαμε την έκθεση αυτή, την δώσαμε στον κύριο Κάρας ακριβώς επειδή είναι πολύ κανός. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να μην μιλήσω τώρα για τα τεχνικά στοιχεία, αλλά για τα πολιτικά. Γιατί θέλουμε την έκθεση αυτή. Φυσικά και μπορεί κανείς να μπει στις λεπτομέρειες, να πει γιατί πρέπει να βελτιωθεί η τραπεζική ρύθμιση, να εκφράσουμε την επιθυμία μας, ότι θέλουμε ακρίβεια. Και όλες οι παρατηρήσεις που γίνανε από αυτού είναι Βεβαίω ενδιαφέρουσε και σωστέ και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. όμω, ποιο είναι ο στρατηγικό στόχο για την έκθεση αυτή. Ο εισηγητή το είπε πάρα πολύ καλά, πιστεύω. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει πρώτα απ' όλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξέρει πριν προταθεί ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί τίνο πρόκειται και ολόκληρη η Ευρώπη πρέπει να τα ξέρει αυτά απέναντι στην Επιτροπή τη Βασιλεία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ποιο είναι το βάρο αυτών που λέμε εμεί σε σχέση με αυτά που κάνει η Επιτροπή Βασιλείας. Ξέρουμε ότι πρόκειται για μια οργάνωση αρκετά κλειστή, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη παρά μόνο τα όσα ενδιαφέρουν εκείνους που συμμετέχουν σε αυτήν. Κατά τα άλλα, ο κίνδυνος που διατρέχουμε είναι να πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην προσαρμογή της οδηγίας μας, να λάβουμε υπόψη αποφάσεις στις οποίες δεν έχει βαρύνει καθόλου δικιά μας η γνώμη. Όμως τα προβλήματα που μας απασχολούν εμάς είναι πρώτα απ' όλα στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Δηλαδή για παράδειγμα ότι στην Ευρώπη παρατηρούμε τα όσα κάνει και λέει η Επιτροπή της Βασιλείας, ενώ η Αμερική καθόλου. Για λόγους τεχνικούς εμείς θεωρούμε ότι μόνο οι τράπεζες διέπονται από τις αρχές της Βασιλείας. Εξάλλου, ο εισηγητή είπε ποια είναι η διαφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Να λοιπόν μια πρώτη στρέβλωση, γιατί οι Ευρωπαϊκέ Τράπεζε τηρούν κανόνε που δεν τηρούν οι Αμερικανικέ τράπεζε. Δεύτερον, το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι θέλοντα να ε, διασφαλίσουμε τι συναλλαγές, βάζουμε ένα σύστημα εγγύσεων για ίδιους πόρους που δεν είναι ρεαλιστικό. Γιατί αν καθίσουμε και κοιτάξουμε τι πρέπει να έχουν οι τράπεζες για να ανταπεξέλθουν ε, στις ρυθμίσεις για τους ίδιους πόρους που σκεφτόμαστε, θα είναι 5 με 6 φορές παραπάνω από αυτά που διαθέτουν σήμερα. Μα τα ποσά αυτά αιτιολογούνται, δικαιολογούνται. Το είπε ο εισηγητής πριν από λίγο, η κρίση από την οποία περάσαμε ήταν μια κρίση ρευστότητας και όχι φερεγγιότητας. Οι τράπεζες δεν ήταν αφαιρέγγες. Η κρίση ξέσπασε στην Ευρώπη, στις τράπεζες, από τη στιγμή που οι τράπεζες δεν είχαν εμπιστοσύνη πια η μία στην άλλη. Και από τη στιγμή που η διατραπεζική αγορά ε, επλήγει. Οπότε τελικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα έπαιρνε από τις τράπεζες και δεν στις άλλες που χρειαζόταν. Λοιπόν, ο εισηγητής πολύ καλά τα λέει. Όλα αυτά διακυδεύονται. Και έτσι. Πρώτον, πρέπει να ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κρατήσει, δεν θα δέχεται οτιδήποτε. Και δεύτερον, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει θέση ανάμεσα στους παρατηρητές της Επιτροπής της Βασιλείας να ξέρει ότι εμείς δεν πρόκειται να εγκρίνουμε το οτιδήποτε. Θέλουμε ασφάλεια στι συναλλαγέ, θέλουμε ισχυρέ τράπεζε, θέλουμε τράπεζε να είναι σε θέση να κάνουν τη δουλειά για τι οποίε έχουν φτιαχτεί, δηλαδή να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη επιχειρήσεων και χωρών, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια ασφυξία στο τραπεζικό σύστημα με απαιτήσει οι οποίε τελικά αποτελούν ψευδέστηση. Θα καταστρέψουμε ακόμη και τι μικρέ τράπεζε, όπω είπατε. Σήμερα λοιπόν αυτό που είναι σημαντικό και πολύ καλά το κάνει ο συγκητής μας είναι να στείλουμε προς τα αυτά τα μηνύματα και να τονίσουμε ότι αν θέλουμε αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα πρέπει να είναι ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο να μπορεί να λειτουργεί και να είναι στην υπηρεσία της οικονομίας και όχι ένα σύστημα ομπρέλας που να προστατεύει αυτούς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ. Έχω δύο γενικές παρατηρήσεις και τέσσερις ε, συγκεκριμένες. Η πρώτη γενική παρατήρηση. Ο στόχος μας με αυτή την γνωμοδότηση είναι να τιμωρήσουμε κερδοσκοπικές συμφωνίες και όχι να δυσκολέψουμε οικονομικές συναλλαγές. αυτή είναι η γενική προσέγγιση και ο γενικός στόχος. Δεύτερη γενική παρατήρηση. Πιο αυστηροί κανονισμοί για τα κεφάλαια πρέπει να εφαρμοστούν και πιστεύω ότι ο εισηγητής έχει δίκαιο το Κοινοβούλιο ενήργησε πιο γρήγορα από ότι η Κομισιόν διότι πιστεύω εμείς ως πολιτικός φορέας αισθανόμαστε περισσότερο την πίεση του χρόνου από ότι η Κομισιόν. Πρέπει να πιέσουμε λοιπόν και την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της. Τώρα οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε τις περιφερειακές επιπτώσεις των κεφαλαϊκών απαιτήσεων. Πρέπει Πρέπει να εξετάσουμε ειδικά τι κάνουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι θηγατρικές τράπεζες. Οι θηγατρικές τράπεζες ε, πολλές φορές ενεργούν ως μοχλή πολιτικής, ε, οικονομικής πολιτικής και επηρεάζουν πάρα πολύ τις εξελίξεις σε μια χώρα που τις ε, φιλοξενεί, στη χώρα υποδοχής. Υποφέρουμε πολλές φορές εμείς από ρευστότητα και δεδομένου ότι θίγονται ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μου, θα πρέπει οι κανονισμοί που διέπουν τις θηγατρικές μεγάλων τραπεζών, να, οι κανονισμοί αυτοί να είναι ακόμα πιο αυστηροί και ε, διαφανείς. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κεντρικών και ανατολικοευρωπαϊκών χωρών και δεν θα πρέπει να δυσκολέψουμε την παροχή δανείων ε, ιδιαίτερα σε μικρότερες επιχειρήσεις και το στραγγαλισμό της ε, ρευστότητας. Οι τράπεζες ε, μας πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν και να εφαρμόσουν τους νέους κανονισμούς και να μην ε, διαταραχθούν ή τελείως σταματήσουν οι διασυνοριακές συναλλαγές, διότι αυτό θα, θα εξαφανίσει τελείως ε, την ρευστότητα. Πρέπει να είμαστε και σαφείς στον ορισμό του βαθμού έκθεσης των τραπεζών σε κινδύνους. Τι εννοούμε ε, έκθεση στον κίνδυνο, ιδιαίτερα στις τράπεζες που κάνουν λιανικές συναλλαγές και σε δάνεια τα οποία δίνονται με ισχύ λιγότερο του ενός έτους η Ουγγαρία έχει εφαρμόσει πολύ αποτελεσματικά μέτρα όσον αφορά τη... την παροχή αυτών των μικροδανείων. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ρευστότητα των θηγατρικών πρέπει να την προσέξουμε ιδιαίτερα. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των στοιχείων σε μια θηγατρική, ακόμα και αν η τράπεζα αυτή είναι ξένη, είναι αλλοδαπή τράπεζα με τη μητρική έδρα σε άλλη επικράτεια. Ε, πρέπει λοιπόν να είναι ε, ανοιχτά τα στοιχεία και προσβάσιμα των θηγατρικών των μεγάλων ξένων τραπεζών Όσον αφορά τώρα το ενεργητικό των, ε, των ε, ταμιευτηρίων θα πρέπει να είναι δημόσια τα κεφάλαια αυτά και να μην εφαρμόζουμε ε, πολύ ε, δύσκολα και άκαμπτα κριτήρια σε αυτές τις ε, τράπεζες. Οι μικρές ε, τράπεζες δεν μπορούν εύκολα να απορροφήσουν κινδύνους και να τους καλύψουν με τα κεφάλαιά τους. Πρέπει λοιπόν να τις βοηθήσουμε. szerintem, nem lehet közvetlenül και επαναλαμβάνω ότι οι μικρές συνεργατικές τράπεζες και τα ταμιευτήρια δεν μπορούν εύκολα να απορροφήσουν μεγάλες ζημιές. Θα πρέπει λοιπόν να τις διευκολύνουμε να διαγράψουν τα ορισμένες απώλειες τους αν μπορούμε όμως να αντικαταστήσουμε τις ζημίες αυτές με την έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι ώστε να δώσουν δυνατότητα και αυτές τις μικρές τράπεζες να έχουν επαρκή κεφαλαϊκά αποθέματα. και να βρούμε ε, τρόπους ε, ε, να εφαρμόσουμε δηλαδή μέτρα τα οποία να είναι αντικυκλικά. Και υπολογίζοντας ε, τα, τα κεφάλαια και κατά πόσο θα είναι η επαρκή πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση ε, πρέπει να χρησιμοποιούμε το κατακεφαλή δίκτυ και να δίνουμε τη δυνατότητα παροχής δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. ευχαριστώ. Εγώ δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα όσα είπαν ήδη συνάδελφοι. Θέλω μόνο να συγχαρώ τον γιατί είναι το θέμα δύσκολο, στόχος της έκθεσης είναι δύσκολο και πιστεύω πως αυτό το κομμάτι είναι, ε, αυτό, ότι αυτή η έκθεση είναι πολύ ισορροπημένη και αποτελεί καλή βάση εργασίας. Θα ήθελα να αναφέρω δύο επιχειρήματα πολιτικού χαρακτήρα, πολιτικής φύσης. Ο στόχος του να εμπλακεί το κοινοβούλιο και να έχουμε μία θέση κινητηρίου δύναμης σε αυτή την υπόθεση νομίζω πως είναι πολύ σημαντικός και από την άλλη πλευρά έχουμε δύο θεμελιώδη προβλήματα. Το ένα είναι ο κίνδυνος ο κλάδος αυτός να πνιγεί θα έλεγα με όλα αυτά που του ζητάμε. Και ως προς αυτό, και εγώ δεν είχα χρόνο να το ψάξω, αλλά ξέρω πως ε, η Τράπεζα Διεθνών ε, ε, Διεθνούς Πύλησης Διαφοράς, Διαφορών ε, International Settlement δημοσίευσε φέτος μια έκθεση και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο αντίκτυπος δεν θα ήταν τόσο πολύ δραματικός όσο εξ αρχής είχαμε πιστέψει με βάση τις πληροφορίες που είχαμε αυτό ότι δηλαδή οι τράπεζες θα πνιγούν από όλες αυτές τις απαιτήσει και αρχίζουν να φαίνονται ε, ε, εργασίες που δείχνουν ότι το μέγεθος αντίκτυπου έχει υπερεκτιμηθεί. Πιστεύω λοιπόν πως αυτά τα έχει ήδη λάβει υπόψη το συνάδελφος Κάρας. Άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η διαφορά των όσων συμβαίνουν εδώ και των όσων συμβαίνουν στην ΕΠΑ. Θα έχουμε μια αντιπροσωπεία την επόμενη εβδομάδα που θα μεταβεί στι ΕΠΑ. Θα μπορούσατε να του ζητήσετε να μεταδιαβιβάσουν τρία-τέσσερα ε, μηνύματα σε σχέση με την κρίση. Η κρίση συνδέεται άμεσα με τα όσα εμείς προσπαθούμε τώρα να ρυθμίσουμε με διαφορετικό τρόπο και άρα λοιπόν θα θέλαμε να στείλει το Κοινοβούλιο ένα μήνυμα και οι διάφορε αντιπροσωπείε που μεταβαίνουν εκεί θα ήθελα να ζητήσω να διαβιβάζουν ένα βασικό θεμελιώδε μήνυμα στου συναδέλφου και στα αμερικανικά θεσμικά όργανα. Αν μπορούσαμε λοιπόν να ρωτήσουμε ποια είναι τα κρίσιμα σημεία αυτού του μηνύματο, θα ήταν πολύ χρήσιμο να τα καθορίσουμε εδώ και έτσι και εμεί να μπορέσουμε όντω να δημιουργήσουμε στην πράξη ένα level playing field, έναν ισότιμο δηλαδή αγώνα με τους εταίρους μας πέραν του Ατλαντικού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γενικώ συγχαρητήρια. Λάβατε κύριε Κάρας, δεν έχω άλλους ομιλητής. Άλλους ομιλητές θέλετε να ολοκληρώσετε. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους σχολίασαν την έκθεσή μου όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους συμφωνούμε όλοι να δώσουμε ένα μήνυμα στην Κομισιόν, ένα μήνυμα στην Επιτροπή της Βασιλείας και να μπορέσουμε τέλος πάντων να ρυθμίσουμε τους δικούς μας ε, κανόνες των δικών μας χρηματοπιστωτικών αγορών. Ξέρουμε ότι εδώ δεν γράφουμε οδηγία, δεν συντάσσουμε οδηγία, αλλά ε, συντάσσουμε μία πολιτική έκθεση και θέλουμε να επηρεάσει αυτή η έκθεση τον τομέα δεδομένου ότι δεν νομοθετούμε. Ένα πολιτικό μήνυμα δίνουμε. Νομίζω ότι και εδώ συμφωνούμε. Τρίτον, όπως η κυρία Φερέιρα είπε, θα είμαι και εγώ μέλος της ε, αντιπροσωπείας που θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να θίξουμε όλα τα ζητήματα αυτά να συζητήσουμε τα αίτια της, κρίσης της κρίσης συγγνώμη, και τα, τις επιπτώσεις εδώ σιγά σιγά έχω την αντίληψη ότι έχουμε προχωρήσει πολύ ήπια μέχρι τώρα. Πρέπει να γίνουμε πιο δυναμικοί. Δεν είναι δυνατόν όλοι να κοιτάνε μόνο το δικό τους το συμφέρον. Πρέπει εμείς εδώ να εκπροσωπήσουμε την Ευρώπη, πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό και είναι απολύτως απαραίτητο να εφαρμόσουμε υπερατλαντικούς μηχανισμούς που να ωφελούν και τις δύο πλευρές. ζητούμε μία έκθεση η οποία να αναλύει τις επιπτώσεις στην πραγματική ζωή, στην πραγματική αγορά. Ε, θέλουμε δηλαδή να φωτίσουμε το σκοτάδι στο οποίο ε, βρισκόμαστε σε πολλές πτυχές. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία λεπτομερέστατη και αναλυτικότατη μελέτη των επιπτώσεων. Όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλια θα, τα, θα τις λάβω υπόψη μου. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θα συνεργαστώ με τη Σκιώδη Συγήτρια και σας παρακαλώ να μου παρουσιάσετε όλα τα, τα ερωτήματα με τα οποία θέλετε να ασχοληθούμε, τα οποία θέλετε να προβάλλουμε και τα οποία να βασίζονται ε, στους πολιτικούς μας στόχους. Διότι ο στόχος της ε, γνωμοδότησης είναι πολιτικός, βασικά. Σας ευχαριστώ κύριε Κάρας. Προθεσμία τροπολογιών 8 Ιουνίου. Θα τη συζητήσουμε στις 28 Ιουνίου και στόχος είναι να ψηφίσουμε στην Επιτροπή 6 Σεπτεμβρίου για την Ολομέλεια 2 του Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Αυτά λοιπόν. Είχαμε να συζητήσουμε το πρωί και θα ξαναρχίσουμε στις 3 η ώρα. Παρακαλώ μην ξεχά... την ηλεκτρονική σας κάρτα, την κάρτα ψηφοφορίας. Έχουμε ακόμα 13 που είναι μέσα στο μηχανάκι.